Okay, we start. No one from the secretary here? No? Okay. Herzlich willkommen. Welcome here. Καλώς ορίσατε. Βλέπετε ότι έχουμε και λουλούδια εδώ μπροστά μας γιατί είναι ιδιαίτερη συνεδρίαση και πολύ όμορφη. Θα ξεκινήσουμε είναι αρκετά φορτωμένη η ημερήσια διάταξη και γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε χωρί καθυστέρηση. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι για την ημερήσια διάταξη. Κατά πόσο εγκρίνεται. Την έχετε μπροστά σα. Να προσθέσω ότι το 17α θα προσταθεί, δηλαδή ανταλλαγή για το COP16. Επί το περιεχομένου το έχουμε διευκρινίσει, αλλά θα θέλαμε να γίνει μια περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. του ζήτησε ο σχετικό συνάδελφο αρμόδιο. Κατά δεύτερον, παρατηρήσει του Προέδρου, ανακοινώσει. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο για το ίδιο θέμα. Ξέρετε ότι εδώ και καιρό, βάσει των ε, διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, συζητήσαμε αναφορικά με το θέμα του COP16 και συμφωνήσαμε ότι θα καταρτήσουμε ε, ψήφισμα. Η κυρία Κορόλα είναι επί της ουσίας ε, αρμόδια. Τους Νόφσκι από Ζαντό, Ματίας, Σαβίνα θα συμμετάσχουν. Κατέληξαν σε συμβιβασμό και το ανέπευσαν το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως είχαμε συμφωνήσει και λογικά έχει συμφωνηθεί το θέμα αυτό, δεν θα πρέπει να δεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία θα γίνει όμως ε, σκεπτική συζήτηση γιατί οι συνάδελφοι θέλουν ε, να σας εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Αυτό θα είναι το 17α της μερίσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλα θέματα και περνάμε... Α, όχι. Δεν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Τι πρόβλημα υπάρχει. Θα μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα σχεδόν προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη. Ξέρετε ότι στη συζήτηση αυτή είχαμε κάνει διάφορες επιμέρους συζητήσεις, αλλά την προηγούμενη φορά είχαμε ε, χρονικούς περιορισμούς. Και επειδή είχαμε αυτούς τους χρονικούς περιορισμούς, είχαμε πει στην συνάδελφο Μπομπίνσκα αν θα μπορούσαμε να ε, βάλουμε το θέμα εκ νέου στην ημερήσια διάταξη για να το ξανασυζητήσουμε. Το βάλαμε λοιπόν ως πρώτο θέμα για να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Αφετέρου, όλοι γνωρίζετε ότι εκ παραλίλου διεξάγονται συζητήσει μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, αφενός και αφετέρου. μεταξύ των ειδικών για το πότε θα οριστεί η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Γιατί ξέρετε, τώρα είναι πραγματικά πολύ άριθμες στον αριθμό αυτέ τις τροπολογίες και αυτό αποδεικνύει άλλωστε πόσο ενδιέφερε το θέμα αυτό του συνοδέλφους, πόσο ενδιέφεραν οι προτάσει σας. Και η κυρία Μπουλίσκα προσπάθησε να τα συνδυάσει όλα αυτά και να συγκεντρώσει τις τροπολογίες αυτές ε, σε κάποιες ομάδες προκειμένου να μην είναι εκατοντάδε ε, στον αριθμό οι, ψηφ... οι τροπολογίε οι οποίε θα πρέπει να ψηφιστούν. Δεν θα το καταφέρει φυσικά για όλε τι τροπολογίε αυτό. Θα πρέπει να ψηφιστούν και κάποιε τροπολογίε. Ωστόσο, βρίσκεται στη διαδικασία σύναψη ε, συμφωνιών. Ναι, αφού κάθισε και συνάδελφο και επειδή μίλησα και αρκετά, να δώσω το λόγο στη συνάδελφο για να μας ενημερώσει να δούμε τι γίνεται με την πρόταση αυτή. Επί του περιεχομένου υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχουν παρατηρήσεις και επί της διαδικασίας, αλλά ας δώσουμε πρώτο λόγο στη συνάδελφο. Thank you very much um, for your kind... Ευχαριστώ για την ευγενική εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε. Um, concerning... Υπήρξε κάποια σύγχυση ως προς το ότι θα γίνουν κάποια σχόλια για το χρονοδιάγραμμα. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει κατεπίγουσα διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να λάβει υπόψη την γνωμοδότησή μας, την έκθεσή μας, στην διαμόρφωση της ενεργειακής της στρατηγικής. Παρόλο όμως που κάναμε ό,τι μπορούμε για να σπεύσουμε και να ετοιμάσουμε την έκθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τελικά δεν τα καταφέραμε και η έκθεση θα περάσει στην Ολομέλεια μετά την έγκριση της στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα δώσουμε την εντύπωση ότι ό,τι και να πούμε για ένα σημαντικό θέμα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θα εγκριθεί εκ των υστέρων η δική μας έκθεση. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ευελπιστώ ότι θα το λύσουμε, ότι η Επιτροπή θα ε, δεχτεί την έκθεσή μας 12 ώρες μετά την συζήτηση στην Επιτροπή την αρμόδια Επιτροπή, τη δική μας. Και εδώ το μήνυμα που θα δώσουμε θα είναι ότι ούτε η Επιτροπή μας, ούτε το Κοινοβούλιο λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά δεν θέλουμε να δώσουμε μια τέτοια εντύπωση. Ελπίζω να καταφέρουμε να το διευθετήσουμε αυτό το πρόβλημα. Όπως ξέρετε, κατατέθηκαν 428 τροπολογίες. Δηλαδή περίπου 10 τροπολογίες για κάθε παράγραφο. Οπότε ουσιαστικά και κάθε παράγραφος της έκθεσης είναι καρπός συμβαστικής ε, πρότασης. Γι' αυτό και εκλυπαρώ την κατανόησή σας. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κάθε συμβαστική πρόταση να καλύπτει πλήρως ε, τις τροπολογίες. Προσπαθούμε να καλύψουμε το νόημα τουλάχιστον, τις βασικές ιδέες. Άλλωστε και οι συμβαστικές τροπολογίες πρέπει να είναι βανάγνωστες και κατανοητές. Γιατί καταρτίζουμε εκθέσεις που δεν είναι για να τι διαβάζουμε μόνο εμεί οι ίδιοι οι ειδικοί, πρέπει να είναι ευανάγνωστες και κατανοητές και για το ευρύ κοινό. Ήδη έγινε ένας γύρος συζητήσεων με τους πιο και οι συζητήσεις αυτές ήταν πολύ επικοδομητικές και ελπιδοφόρες για την έκβαση της έκθεσης. Μόλις μια εβδομάδα μας έχει απομείνει για να ολοκληρώσουμε την κατάρτιση των συμβαστικών ε, τροπολογιών, ελάχιστο χρόνο δηλαδή, γιατί μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να έχουμε καταλήξει στις συμβαστικές προτάσεις. Ελάχιστα σημεία έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή που να είναι όντως επίμαχα και να υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων. Θα επιχειρήσουμε βέβαια συμβαστικές ε, τροπολογίες και για αυτά τα επίμαχα σημεία, αλλά μπορεί και να μην θα καταφέρουμε, οπότε θα πρέπει να ψηφιστούν ξεχωριστά. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας είναι ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα, γιατί φυσικά υπάρχει διάσταση απόψεων και εντός των κομμάτων. Και στο ΕΛΚ έχουμε διαφορές και σε άλλες ομάδες. Γι' αυτό και θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας. Ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Δεύτερο ζήτημα, αρκετά επίμαχο, είναι η δεσμευτική, υποχρεωτική στόχη για την ενεργειακή αποδοτικότητα μερικές χώρες είναι πολύ απρόθυμες με τον υποχρεωτικό αυτό χαρακτήρα. Το θέμα συζητήθηκε κτένος και έχω την αίσθηση ότι όλες οι σχετικές τροπολογίες για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των στόχων της ενεργειακής αποδοτικότητας θα πρέπει να μεταφερθούν στην έκθεση Benson. που θα συζητηθεί σχεδόν παράλληλα με τη δική μου έκθεση. Η έκθεση Μπένσον είναι πιο κατάλληλη για τα θέματα αυτά γιατί αφορά ακριβώ την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα σα έλεγα λοιπόν να αφήσω αυτή τη συζήτηση εκτό του πεδίου τη έκθεσή μου. Τα θέματα των υποχρεωτικών στόχων, δεσμευτικών στόχων, να το αφήσουμε για την έκθεση Μπένσον. Δεν θέλω να μεταφέρω δηλαδή, τα επιμάχα σημεία αλλού. Αλλά θα έχουμε ένα δεκαετές πρόγραμμα για την ενέργεια. Αυτό είναι το θέμα της έκθεσής μου και καλό θα είναι να περιοριζόμαστε σε αδρές κατευθυντήριες γραμμές και να μην επισέλθουμε σε σημαντικά μεν, αλλά πολύ πιο ειδικά ζητήματα. Θα έλεγα να μείνουμε στα πιο γενικά θέματα προσανατολισμού στη δική μου έκθεση. Ένα άλλο ακαθόδε ζήτημα είναι η χρηματοδότηση. Η ενέργεια είναι ένας κλάδος που δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Ούτε προσελκύει αρκετά επενδυτικά κονδύλια. Χρειάζεται σημαντική οικονομική στήριξη. Βέβαια, ο καθένα ζητάει χρηματοδότηση συγκεκριμένου θέματο ή προγράμματο. Αλλά δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για να ικανοποιηθούν όλοι. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο διορατικοί και να έχουμε πιο μακροπρόθεσμους στόχους στο θέμα της ε, χρηματοδότησης. Ε, εγώ είμαι υπέρ της πρότασης Μπούζεκ, γιατί από τη στιγμή που μιλούμε για κοινέ αγορές ε, και κοινοτικέ μεθόδους στην ενέργεια, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, ομάδες ε, αγοράς όπως αυτή που προτάθηκε για το φυσικό αέριο. Γιατί τέτοιου είδου ομάδε μπορεί να είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση και να πετύχουν καλύτερε προσφορέ από ό,τι μονομένε χώρε. Αλλά βέβαια δεν είναι τη αρισκία όλων αυτό το θέμα. Θέλω να μου πείτε τις απόψεις σας. Και ο κύριος Βόμποντα το πρότεινε. Όπως σας είπα, στις συμβαστικές προτάσεις θα προσπαθήσω να καλύψω όσο το δυνατό περισσότερες τροπολογίες γίνεται. Και υπάρχουν αρκετές και ενδιαφέρουσες τροπολογίες για πολλά θέματα. Εγώ προσπάθησα πολλές παραγράφους να τις συμπτύξω σε γενικές παραγράφους. Υπάρχουν πολλές τέτοιες γενικές παραγράφοι που καλύπτουν περισσότερες τροπολογίες. Θα δούμε τώρα ποιες τροπολογίες ε, θα γίνουν δεκτές αυτούσιες, ποιες ε, καλό θα ήταν να αποσυρθούν. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμη για να τελειοποιήσουμε τις προτάσεις μας και τους συμβιβασμούς και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως τους συμβούλους, βοηθούς και τη γραμματεία που κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτό το πολύ φορτωμένο και πιεσμένο χρονοδιάγραμμα που έχουμε και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί πραγματικά του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τις ε, πληροφορίε που μας δώσατε, αλλά και κατά δεύτερο λόγο για τη δουλειά σα, η οποία έλαβε χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκε. Ο κύριος Ρόντε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπομπίνσκα για έναν πολύ ειλικρινή τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό, με τόσες πολλές τροπολογίες, αλλά πραγματικά μέχρι τώρα έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε όλες, όλες τις προσωπικές μας προτεραιότητες, αλλά διαβάζοντας τις τροπολογίες, νομίζω ότι η προοπτική συμβιβασμού των τροπολογιών ε, είναι αρκετά καλή. Για μας η χρηματοδότηση, η έρευνα, η ανάπτυξη, η εστίαση στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν να είναι βασική προτεραιότητα. Θα ήθελα επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ο οικονομικός ε, αντίκτυπος ε, της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν με απασχολεί. Δεν θα μιλήσω τόσο για την ουσία της έκθεσης, γιατί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με αυτό. Όμως, η Επιτροπή ανακοίνωσε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα και αυτό με ανησυχεί. Και το είπε και η κυρία Μπομπίνσκα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε το χρονοδιάγραμμα. αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω. θα παρουσιάσει την ενεργειακή πολιτική στις 27 Οκτωβρίου. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Αν ισχύει ωστόσο αυτό, προτείνω ο Πρόεδρος να αποστείλει επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διευκρινίσει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποτεκτό ούτε από την Επιτροπή μας, ούτε από το σύνολο του Κοινοβουλίου. Ίσως όμως θα μπορούσε να διευκρινίσει ο Πρόεδρος αυτό άμεσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφε. Να προσπαθήσω να απαντήσω καταρχάς. Έγινε μια τέτοια συζήτηση στο Στρασβούργο. Συνεμίλησα με την Επίτροπο και μου είπε ότι αυτό θα συμβεί στις 3 Νοεμβρίου. Αυτό είναι γεγονός. Βελτιώθηκε λοιπόν κάπως η κατάσταση και χτες ακούσαμε αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ότι προβλέπετε στις 27 Οκτωβρίου στην ημερήσια διάταξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ θεώρησα ότι αυτό είναι απαράδεκτο, όπως και εσείς άλλωστε, γιατί όταν έχουμε κάτι συμφωνήσει, το έχουμε συμφωνήσει και το ρώτησα γραπτά και με ενημέρωσαν χτες, χτες το βράδυ από το γραφείο του κ. Ότιγκερ ότι πρέπει να μπει στις 27 Οκτωβρίου γιατί στις 3 Νοεμβρίου είναι πράσινη εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα δημοσιευτεί αργότερα, πολύ αργότερα, στις 9 του μηνός. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Σε περίπτωση που φυσικά αλλάξει αυτό, θα πρέπει αυτό να μας επηρεάσει και εμάς, να προσαρμόσουμε και εμεί την τρόπο εργασία μας και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί έχουμε χρονικού περιορισμού ήδη για αρχές Νοεμβρίου. Ε, και εγώ αναμένω ότι θα τηρηθούν οι υποσχέσεις αυτές. Σε περίπτωση που υπάρχει τώρα εκ νέου αλλαγή, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, αλλά φυσικά θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τη δικιά μας ψηφοφορία στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα, κυρία Τζαβέλα. Και σκιώδης και αυτή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα, με τους συναδέλφους κύριε Μπούτι, κύριοι, ε, κυρίους Μπούτι Κόφερ και Τσουκαλά, έχουμε προτείνει ε, ένα νέο recital. Αλλά πριν πω σε αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ την συγγραφέα της ε, ε, αναφοράς, την κυρία Μπομπίνσκα, εξαιρετική δουλειά για μια πολύ σημαντική και στρατηγική πράγματι ε, εργασία για την ε, Ένωση και τους πολίτες της. Κυρία Μπομπίνσκα, τα συγχαρητήριά μου και μπαίνω στις προτάσεις μας. Με τον κύριο Μπούτι Κόφερ και τον κύριο Τουκαλά έχουμε βάλει ένα καινούριο recital το οποίο υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρόθεση που είχε εκφράσει η Επιτροπή στο παρελθόν για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για το LNG. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο προτείνουμε να μπει ως recital. Στην παράγραφο 4, <clears throat> για ορθολογικούς λόγους, έχουμε βάλει τη λέξη μεσοπρόθεσμα, δηλαδή υπάρχει ε, ο χαρακτηρισμός βραχυπρόθεσμα action plans και θα λέγαμε για ορθολογικούς λόγους να βάζαμε και το μεσοπρόθεσμα για να είμαστε πιο ε, συνεπείς με ένα πρόγραμμα το οποίο θα κυλήσει. Στην παράγραφο 28, προς το τέλος, ενώ το κείμενο αναφέρεται σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για την ε, περιφερειακή αγορά των ανανεώσιμων πηγών. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να είμαι αρκετά ρεαλιστική. Θα έλεγα ότι είναι μακροπρόθεσμο αυτό παρά μεσοπρόθεσμο. Δηλαδή, σε πολλά κείμενά μας θα πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα για να επιτύχουμε μια περιφερειακή αγορά ανανεώσιμων πηγών. Δεν νομίζω ότι θα γίνει μεσοπρόθεσμα. Χρειάζεται πολλής χρόνος και θα ήμασταν πολύ ρεαλιστέ αν αντί για το μεσοπρόθεσμο αναφερόμασταν σε μια μα, ε, μακροπρόθεσμη ε, χρονική διάρκεια. Ε, η τελευταία ε, προσθήκη που θα ήθελα να κάνω είναι στην παράγραφο 32. Εδώ προτείνω την επέκταση της ενεργειακής κοινότητας σε τρίτες χώρες που είναι και προμηθευτές όπως ο κόλπος και η Μέση Ανατολή. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους κυρίους συναδέλφους και σε εσά κύριε Πρόεδρε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο Επίτροπος κύριος Ότιγκερ στην Ολομέλειά μας επιβεβαίωσε ρητά ότι θα δοθεί έμφαση στις χώρες που είναι και παραγωγή ενέργειας, ανέφερε δε όπως η Μέση Ανατολή και το Κατάρ. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω στην παράγραφο 32 να δεχθείτε την ε, ε, πρόταση την οποία έχω διατυπώσει ως επέκταση της ενεργειακής κοινότητας σε τρίτες χώρες που είναι παραγωγή ενέργειας, Μέση Ανατολή και Κόλπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γκουρκ γιατί την προηγούμενη φορά συμφωνήσαμε όσοι είχαν μπει στον κατάλογο μιλτών να πάρουν πρώτοι το λόγο. Συνάδελφε, έχετε το λόγο και μετά οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά δύο στοιχεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. Αν ε, συνεχίσει με τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει... Τι, τι θα γίνει, θα γίνει τεχνική συνεδρίαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα παίξει το ρόλο που θα πρέπει να παίζει. Και θα έπρεπε πραγματικά να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα τέτοιο στρατηγικό θέμα. Το δεύτερο στοιχείο με το οποίο πρέπει να συμφωνήσω είναι το εξή. Η συγγήτρια όντω δυσκολεύτηκε πάρα πολύ εν ώψη και του όγκου που καλύπτει το θέμα, αλλά και των ε, πολυάριθμων τροπολογιών. Καταλαβαίνω αυτά που λέει η συγγήτρια ότι θα ήθελε να μπορούσαν να αποσυρθούν κάποιες ε, οι τροπολογίες. Αυτό θα τη βοηθούσε ιδιαίτερα. Εγώ ωστόσο δεν θα το πράξω αυτό. Θα προτιμήσω να τη βοηθήσω υποστηρίζοντας τις τροπολογίες που υπέβαλα. Θα ήθελα να θίξω τέσσερα θέματα. Καταρχάς, η δημιουργία θέσεων εργασίας. Σωστά, πολύ σωστά επιμένει η έκθεση για τη διασφάλιση περαιτέρω κονδυλίων για την επόμενη χρηματοοικονομική περίοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο πολλοί πόροι για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Το σχέδιο της ανάκαψης της οικονομίας δεν ήταν αυτό που θα επιθυμούσαμε. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το βελτιώσουμε αυτό. Και όταν μιλάμε για την ανάκαμψη της οικονομίας και τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, θα πρέπει πάντα να μην ξεχνάμε την πτυχή της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε καμία περίπτωση. Δεύτερο θέμα, επενδύσεις. Αυτό που είναι θετικό στην έκθεση είναι ότι είναι πάρα πολύ γενναίος ο τρόπος με τον οποίο ονομαστικά αναφέρονται επενδύσεις. Για παράδειγμα, το Ναμπούκο. Συμφωνούμε με την αναφορά αυτή, αλλά θεωρώ ότι κατά τη δεύτερη εξέταση οι στόχοι που έχουμε θέσει δεν έχουν χάσει τίποτα από την αξία τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια, κάποιους στόχους εκτός, γιατί και αυτό θα αποτελούσε μήνυμα, αν θέλετε. Να αναφέρουμε λοιπόν συγκεκριμένα, ονομαστικά κάποια θέματα για τα LNG, για την ε, Μεσόγειο, το αέριο, τους διασυνδέσεις, το δίκτυο offshore της Βόρειας Θάλασσας. Φυσικά δεν πρέπει να φορτώσουμε περιτά την έκθεση, αλλά να μην περικόψουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν θα εξαρτηθεί από αυτό το μέγεθος και η έκταση της έκθεσης. Τρίτο θέμα. Τα κίνητρα που θα δοθούν στην αγορά. Είναι σημαντικό οι πόροι να διευρυνθούν. Συμφωνώ με την υποστήριξη των επενδύσεων, αλλά δεν θα αρκέσουν οι κοινωτικοί πόροι. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τα κίνητρα της αγοράς. Θα πρέπει να ορίσουμε ως στόχο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εναρμονίσουν τα κίνητρα προς τον ενεργειακό τομέα, είτε με φορολογικούς τρόπους, είτε με άλλους τρόπους. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεστική λειτουργία της αγοράς. Τέταρτο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, οι ανανεώσιμες και τα θέματα ιδιαίτερα της έγκρισης, της αδειοδότησης των ανανεώσιμων. Φυσικά δεν είναι στόχος της έκθεσης να εστιαστεί αναλυτικά σε θέματα αντιεδότησης των ανανεώσιμων. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά θεωρώ ότι στο κεφάλαιο για την ενεργειακή ασφάλεια θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη σημασία οι ανανεώσιμες. Γιατί όντω μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μείωσης της ε, εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ξένες εισαγόμενες ενέργειες θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εναρμονίσουν τις πτυχές που αφορούν την αδειοδότηση τις ε, ανανεώσιμες και θα πρέπει να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές μέχρι το 2020 και αυτό το λέω ως ε, εκπρόσωπος μιας χώρας η οποία χρειάζεται 40 με 50 άδειες ε, ανανεώσιμων προκειμένου να φτάσει σε ένα σωστό επίπεδο. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να αναφέρω που αφορούν τις τροπολογίες μου και ελπίζω να προσθεθούν αυτά τα θέματα στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος ένας κοιόδης, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσουμάνσκι. Θα του δώσω πρώτο το λόγο επειδή είναι ε, κοιόδης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τον ε, προηγούμενο μιλητή. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους ε, εξάφρασαν τη δυσαρέσκειά τους γιατί είναι πολύ πιθανόν η έκθεσή μας τελικά να μην έχει καμία απολύτως επιρροή στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ εγκαίρως στις εργασίες μας πριν από την ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελικά δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Πολύ άριθμες ήταν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν και πάρα πολλοί βουλευτοί θέλουν, βουλευτές συγγνώμη, θέλουν να επηρεάσουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ λοιπόν τον πρόεδρό μας να τηρηθούν οι ανάλογες προθεσμίες για να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια καλή αρχή. Η ομάδα μας υπέβαλε πάρα πολλές τροπολογίες και θεωρώ ότι πολλοί είναι και οι συμβασμοί οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν. Το θέμα είναι να υπάρξουν συμφωνίες χρήστη. Να δούμε δηλαδή συμφωνίες οι οποίες στο μέλλον θα ωφελήσουν τον πολίτη η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών είναι απαραίτητη, γιατί αυτό φυσικά είναι ευεργητικό για τον ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός είναι σημαντικό στοιχείο για μας και για το χρήστη και κάτι ακόμα θετικό είναι οι δυνατότητες της ε, πυρηνικής ενέργειας. Δεν μιλάμε μόνο για χαμηλή χαμηλό ποσοστό α, ρήπων. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα τις εργασίες μας προκειμένου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος Κάριντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω συγχαίροντας τη συνάδελφο Μπομπίνσκα για μια πολύ καλή δουλειά. Είναι γεγονός ότι συχνά λέμε συγχαρητήρια, αλλά μερικές εκθέσεις το αξίζουν περισσότερο. Μας δίνει σαφείς επιλογές ε, η συγκίδρια. Θα ήθελα όμως μία πτυχή ιδιαίτερα να τονίσω και αυτή είναι η σημασία Τη ολοκλήρωση των διασυνδέσεων ε, προκειμένου να υπάρχει ένα ε, διαδίκτυο και στην αγορά ηλεκτρισμού και στην αγορά ε, αερίου. Υπάρχει το θέμα της απομόνωσης ορισμένων χωρών από τις αγορές αυτές. Αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του, αλλά πιο σημαντικό ακόμα όταν σκεφτόμαστε στο πλαίσιο της κρίσης και όταν σκεφτόμαστε κυρίως τι νομοθεσία θα μπορούσαμε να έχουμε προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στα κράτη-μέλη, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι η ενίσχυση ε, του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, γιατί μεγαλύτερος ε, ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων, μειώνει τις τιμές για τους καταναλωτές και φυσικά δεν διαφέρει σε τίποτε αυτό η ενέργεια, γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κινηθούμε προς ε, μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε και ενιαία δίκτυα με σκοπό να έχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στις χαμηλότερες τιμές προς τους τελικούς καταναλωτές. Και η έκθεση αυτή αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα σε πολλά σημεία Νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε το θέμα αυτό και να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη ίδρυσης δικτύων, ώστε να υπάρχουν οι συνθήκες μιας ανοιχτής αγοράς ενέργειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. πολύ δύσκολο το εγχείρημα της κυρίας Μπομπίνσκα. Όχι μόνο επειδή είναι ίδιας πρωτοβουλίας, αλλά επειδή όλα τα θέματα τα εξετάσαμε στα πλαίσια του σχεδίου έκθεσης. Γιατί είναι σαν να, έχουμε, να αμφισβητούμε κάτι που στο παρελθόν είχαμε εγκρίνει, σαν να είναι ψήφος μορφής προς αυτά που προς το παρελθόν εγκρίναμε. Βέβαια, άλλο θεωρία και άλλο πράξη. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πακέτο, είπαμε ότι ο άνθρακας και στο μέλλον θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενέργεια, στο ενεργειακό πακέτο. Ενώ αυτό το πακέτο φαίνεται ότι μπλοκάρει την ενέργεια με βάση τον άνθρακα ως βασική πρωτήλη. Ενώ η βιομηχανία που στηρίζεται στον άνθρακα δεν θα πρέπει να υποστηρίζεται μόνο από μονομένες τεχνολογικές μεθόδους όπως είναι δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, αλλά θα πρέπει να ε, ενισχύεται. Οπότε οι λεπτομέρειες θα πρέπει να περιληφθούν στο δεύτερο σχέδιο του κυρίου Μπέντ αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και εδώ και για την ε, ε, γενική αποδοτικότητα. Επίσης, στο θέμα συμπαραγωγής ενέργειας, κατά 80%. Γιατί αν οι νέοι ηλεκτρικοί σταθμοί με βάση την, ε, τον άνθρακα έχουν καλύτερου τρόπου για την αποθήκευση του άνθρακα, αυτό θα πρέπει να ισχύει, αν έχουμε τέτοιε απαιτήσει από τον άνθρακα, να ισχύει και από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με άλλα μέσα, όπως με το πετρέλαιο για παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τέτοιου είδους ε, τροπολογίες. Γιατί δεν είναι νομοθετικό αυτό το σχέδιο. Θα πρέπει να δώσουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να μην ξεχνούμε και το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πακέτο. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ήδη εγκρίνουμε αυτό το ενεργειακό περιβαλλοντικό πακέτο υπό την ε, ε, επιρροή των πρασίνων κυρίως που μας είχαν πείσει ότι το COP15 είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει η Ευρώπη να αποδείξει στον κόσμο πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ήρθε όμως το μεταξύ η οικονομική κρίση και, και η ενεργειακή κρίση και μας έδειξε πόσο σημαντική είναι και η ενεργειακή κρίση για μια οικονομία που στηρίζεται στον άνθρακα, όπως είναι η οικονομία της Πολωνίας, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο Φόγκοντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο, η συγγήτρια, για την εργασία της να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είναι δύσκολο να καταρτιστεί μια γενική στρατηγική όταν ε, προστίθενται πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες εκπροσωπούν μονομένα συμφέροντα και συμφωνώ με τη συνάδελφο ότι δίκαιο έχει το πιο σωστό θα ήταν να προσταθούν αυτά τα μονομένα θέματα σε ό,τι αφορά τους μεμονωμένους και ξεχωριστούς νόμους. Να πω επίσης ότι επί της αρχής ε, συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε μια οικονομία χαμηλή σε εκπομπές άνθρακα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τεθούν κάποια σημεία προτεραιότητας και θα θέλαμε στην Αυστρία για παράδειγμα να θέσουμε το θέμα της ε, υδροελεκτρικής ενέργειας. Μία παρατήρηση να κάνω για τις χρηματοπιστωτικές ε, αγορές, επειδή το είπε και στον άδελφος. Σωστό είναι να ζητάμε ε, ευρωπαϊκά κονδύλια για τις ε, υποδομές. Αλλά το θέμα είναι, θέλουμε να υπάρχει επιρροή της ομάδας μας. Θα πρέπει να γίνει σχετικός αγώνας για το, τους πόρους αυτούς και τον υπερπολογισμό σε όλες τις ε, επιτροπές. Ακούω για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση της Ολλανδίας των κατοχωρών θέλει να μειώσει στο ίμιση της ε, τη. της. Άμα ε, ισχύουν αυτά θα πρέπει να ξεχάσουν τα σχέδιά μα. Και τελευταίο σημείο τώρα. Η συνάδελφος Μπομπίνσκα ναι. ανέφερε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε μετά και από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας βλέπουμε ότι όλο και πιο πολλοί εμπειρογνώμονες και πολιτικοί από την, ε, τις εθνικές κυβερνήσεις λένε ότι χρειαζόμαστε πιο, πολύ, πιο πολλές υποδομές. Είτε πρόκειται για δίκτυα, είτε πρόκειται για βιώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός σύνδεσμος προκειμένου να δούμε και τι γίνεται και με τις διαπραγματεύσεις. Είτε μιλάμε για τη Ρωσία, είτε μιλάμε για το Κάφκασο, είτε για μιλάμε για την Κίνα. Όλα συνηγορούν στο ότι θα πρέπει από πλευρά ενεργειακή πολιτική να ενισχύσουμε την Ευρώπη χωρί να γίνουν διαφοροποιήσει μεταξύ των χωρών. Θα πρέπει από κοινού να καταρτήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα είναι παραπάνω από αυτά που ήταν έω τώρα. Μύρισα και με την κυρία Μόντε, τον κύριο Μόντε, ο οποίο ήθελε φυσικά την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγοράς, αλλά είπε ότι άλλοι δεν υποστηρίζουν αυτή την ε, ενιαία αγορά. Στην Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική η οποία θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και αυτό θα συνδεθεί και με την ε, δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις της εταιρεία ε, αερίου, το οποίο επηρεάζει και τις τιμές του αερίου. Και φυσικά αυτό δεν είναι απλό εγχείρημα. Ακούσαμε και τον Επιτροπό που μίλησε για τα πιο πρακτικά προβλήματα και νομίζω ότι με την έκθεση της κυρίας Μπομπίνσκα μπορούμε να αποστείλουμε κάποια σαφή μηνύματα ότι θέλουμε να πετύχουμε πιο πολλά χωρίς να θίξουμε το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας, γιατί νομίζω ότι ήταν αρκετά δύσκολο να πετύχουμε την Λισαβόνα βάσει της σύμβασης αυτής. Είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, το οποίο είναι θετικό. Χαίρομαι που μας υποστηρίζει η κυρία Πομπίνσκα. Και έχουμε συμφωνήσει να συμπεριλάβει τέτοια στοιχεία στην έκθεσή τη, γιατί αυτά τα μηνύματα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις επιμέρου εκθέσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι θα ήθελα να πω ότι σχεδόν όλοι όσοι εργάζονται στον ενεργειακό κλάδο στην Ευρώπη θέλουν όχι πιο λίγα, αλλά πιο πολλά να δουν από τον κλάδο αυτό. Και αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν δεν υπάρχει πιο έντονο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό να μεταφερθεί και προ τα έξω. Ο συνάδελφο Μεσάντης λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετική σημασία ε, αυτή η έκθεση. Εμείς ε, τρει συνάδελφοι έχουμε υποβάλει τρεις ε, ε, πέντε τροπολογίε οι οποίες ελπίζουμε να συμπεριληφθούν. Εκτιμώ ιδιαίτερω τις προσπάθειες της κυρίας Μπομπίνσκα να είναι επιτυχής η έκθεση. Χρειαζόμαστε μία νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία ασφάλεια ανεφοδιασμού, αποδοτικότητα της ενέργειας ε, και κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όταν μιλάμε για ενεργειακή πολιτική, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι δεν δρούμε τόσο για το παρόν όσο για τις μελλοντικέ γενναίες. Επομένως, ε, νέες ε, τεχνολογίες χαμηλής, χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντικές είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ε, συμπεριλάβουμε στη στρατηγική μας. Όχι μόνο οι πρόσφατες τεχνολογίες, όλες οι τεχνολογίες που πρόκειται να αναπτυχθούν, ε, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των ε, πυρηνικών μορφών ενέργειας επίσης. Η ρήτρα της αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στην έκθεση δεν είναι μόνο προ συμφέρον ε, των κρατών μελών, ε, του κάθε κράτου μέλου, ε, όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Ελπίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα Ναμπούκο, μπούκο να διατηρηθεί γιατί θα δώσει τη δυνατότητα αυξημένης ανεξαρτησίας σε σχέση με τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Taip pat e, noriu padėkoti Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Πομπίνσκα για το κείμενο αυτό το οποίο προσανατολίζεται πραγματικά στο μέλλον. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες καταδεικνύει ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση και ότι δεν θα είναι απλό να εξευρεθούν συμβαστικές προτάσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Σβόμουντα που πήρε το λόγο και είπε ότι είναι πλέον ε, καιρός στα θέματα της ενέργειας να υπάρξει πιο πολύ Ευρώπη. Γιατί συχνά έχουμε διαφωνίες επί σειρά ετών για θέματα, αλλά κάποτε θα πρέπει να ακολουθήσουν και πράξεις. Δυστυχώς, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής δεν είχαμε χρόνο, γιατί ήθελα να πάρω το λόγο και τότε. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τη σύμβαση μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας σε ό,τι αφορά την συνέχιση των εκμεταλλεύσεων μέχρι το 2000 Πρόκειται δηλαδή για όρους οι οποίοι έχουν τεθεί και οι οποίοι θα ισχύουν για 35 χρόνια. Αυτό ανταποκρίνεται με τις στρατηγικές μας. Είναι σωστό. Θα ήταν δυνατόν με τον τρόπο αυτό να καταρτιστεί στρατηγική, να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές πηγές και οι σωστές τιμές. Νομίζω ότι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμειγνύεται σε τέτοιες ε, συμφωνίες δεν είναι πλέον επίκαιρο, δεν είναι πλέον σωστό για το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Και συμφωνώ και με τους συναδέλφους που είπαν ότι είναι σημαντικό να συνδεθούν οι ενεργειακές ε, νήσοι. Θεωρώ λοιπόν ότι η τροπολογία 4 θα πρέπει να παραμείνει στην έκθεση αυτή. Εμείς ε, ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμείνουμε στη θέση μας. Συμφωνούμε επί των πλέον σημαντικών πτυχών σε ό,τι αφορά την αγορά αερίου. Εντάξει, συμφωνούμε, πρόκειται για ένα πρώτο βήμα στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές εκτός της Ένωσης. Πιστεύω ότι στις εργασίες ε, της ομάδας αυτής ε, αγοράς θα πρέπει να διευκρινίζουμε σημαντικά θέματα, τα οποία θα καθορίσουν την στρατηγική. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Αν συμφωνείτε, επειδή έχουν ζητήσει το λόγο άλλοι οκτώ ομιλητέ, θα ήθελα να κλείσω στο σημείο αυτό το κατάλογο των ομιλητών. Αν δεν έχετε αντίρρηση, ο συνάδελφο Κουάντρα. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Κολάρσκα Κολάρσκα-Βομπίνσκα γιατί μας παρουσίασε μια έκθεση που έχει μια σημαντική αρετή. Είναι πλήρης, ισορροπημένη και λογική η έκθεσή της. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν την έκθεση ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας. Αν θέλουμε ως κοινοβούλιο, κίτρε, να τα καταφέρουμε, θα πρέπει να αποφύγουμε ε, τροπολογίες που είναι άσχετες με το κείμενο της κυρίας Κολάσκα Μπομπίνσκα, που όπως είπα είναι αρκετά ισορροπημένο. Εγώ κατέθεσα αρκετές τροπολογίες που αυτή τη γραμμή ακολουθούν, αυτή την κατέθεση, Δηλαδή, βελτιώνουν κατά τη γνώμη μου το κείμενο, αλλά δεν το τροποποιούν άρδιν. Ούτε παραμορφώνουν ούτε αλλοιώνουν την έκθεση της κυρίας Κολάρσκα όπως επιχειρούν άλλες τροπολογίες. Γιατί κατά τη γνώμη μου τέτοιου είδους τροπολογίες θα ήταν λάθος να γίνουν δεκτές. Από τις πολυάριθμες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί δημιουργείται πρόβλημα με εκείνες τις τροπολογίες που είτε εκπορεύονται από υπερβολικά εθνικιστικές ιδεολογίες ε, συμφέροντα, είτε ε, τις τροπολογίες που εμπνέονται από πολύ ουτοπικές φιλοδοξίες. Επίσης πρόβλημα υπάρχει με ορισμένες τροπολογίες που είναι άσχετες ε, και προτάσεις που είναι άσχετες με το πεδίο εφαρμογής αυτής της έκθεσης. Είναι εκτός θέματος ουσιαστικά οι τροπολογίες αυτές. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή μας έχει δείξει σοβαρότητα, ρεαλισμό, υπευθυνότητα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε με την κυρία Κολάρσκα, να καταλήξουμε σε συνετές συμβαστικέ λύσεις, όλοι να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις για να κερδίσουμε και ορισμένα από τα σημεία που μας ενδιαφέρουν και να αποφύγουμε είτε τις υπερβολικά ε, εθνοκεντρικές ε, προσεγγίσεις είτε τις υπερβολικά ουτοπικές απαιτήσει. Η έκθεση αυτή είναι πολύ εύστοχη γιατί καθορίζει κάποιες στρατηγικές καταθεντήρες γραμμές για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτούς τους προσανατολισμούς που προτείνω, τα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρα στο έργο μας. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Μπομπίνσκα για τη δουλειά της. Να της ευχηθώ καλό κουράγιο σε σχέση με την χιονοστιβάδα τροπολογιών που υπευλήθησαν. Πρόκειται για κάτι που το συζητούμε πολλά χρόνια και το γεγονός ότι έχουμε αυτή την έκθεση το αποδεικνύει. Η νέα στρατηγική ενέργειας πρέπει επίσης να έχει μια, ένα κοινωνικό περιεχόμενο, μια κοινωνική πτυχή. Πάνω από 50 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίοι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ε, τους λογαριασμούς ε, ενέργειας. Πρόκειται για κάτι που, είναι, που πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και ειδικότερα στην έκθεση αυτή γιατί η στρατηγική 2003 με 2009 περιείχε μία ρήτρα υποχρεωτικής ε, ε, πρόβλεψης ε, χαμηλότερων τιμών για αυτούς που βρίσκονται σε, πιο, σε λιγότερο καλή οικονομική κατάσταση. Οι Υπουργοί Ενέργειας που συνεδρίασαν το Σεπτέμβρη ζήτησαν εθνικές λύσεις ε, και παρέπεψαν το θέμα στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι πρέπει να παρέμβουμε και να επηρεάσουμε την κατάσταση. Ναι, μεν πρέπει να υπάρξουν εθνικοί στόχοι για την ε, μείωση της φτώχειας, αλλά πρέπει να έχουμε και μία στρατηγική. Και το λέω αυτό ε, και σε σχέση με όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι μέχρι τώρα. Πρέπει να κινηθούμε προς μια πραγματική ε, ενεργειακή κοινότητα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, για την διαδικασία συζητάμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μία προσέγγιση ότι λυπούμεθα για λογαριασμό τους, γιατί δεν έχουν, δει, δεν έχουν καταλάβει καθόλου την άποψη του Κοινοβουλίου ως προς αυτά τα ζητήματα και στο τέλος, όταν ε, υπάρχει νομοθεσία, όταν πρόκειται για νομοθεσία, οι αποφάσεις θα ληφθούν εδώ θα είμαστε αυστηροί, κατηγορηματικοί όταν παρουσιάζουμε ε, πράγματα που για μας είναι σημεία αφετηρίας. Δεύτερος προβληματισμός σε σχέση με την ουσία. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση της εισηγήτριας, την οποία θα ήθελα και να συγχαρώ, γιατί είναι μια πολύ καλή έκθεση. Τα δίκτυα, ε, η διασύνδεση είναι πραγματική, είναι πραγματική όροι προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, τους στόχους μας. Ε, δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε τίποτε χωρίς να έχουμε καλύτερη ε, λειτουργία των δικτύων, των ευρωπαϊκών δικτύων. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο. Και επειδή αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ε, εφαρμογή της εξωτερικής πτυχής ε, της ενεργειακής ε, πολιτικής και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νομίζω ότι το σχέδιο Ναμπούκο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Να τονίσουμε επίσης την ανάγκη έμφασης στις σημαντικότερες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα της πυρηνικής ενέργειας είναι ένα τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και ότι θα έχουμε κλιματικώς ε, ευφυή παραγωγή ενέργειας. Και δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό χωρίς να τονίσουμε την ανάγκη ύπαρξης ε, πυρηνικής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και λυπούμε και την καθυστέρηση. Θερμά ευχαριστώ στην κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα γιατί είναι τεράστιο αυτό το εγχείρημα της προσπάθειας συμπίλησης 500 σχεδόν τροπολογιών. Και οι συμβαστικές τροπολογίες που μας έστειλε χθες το απόγευμα είναι πολύ καλή βάση και σημείο αφετηρίας για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Τώρα επανέρχομαι στο θέμα του χρονοδιαγράμματος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι προκλητική η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπή δεν έχει κανένα, καμία ανάγκη να ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη μέσα Οκτωβρίου και τέλη Νοεμβρίου να αφήσει το θέμα για έγκριση, πάλι προλαβαίνει να το υποβάλει στο Συμβουλίο Υπουργών. Γιατί αυτή η βιασύνη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία παρατήρηση, το εξηγήσαμε στην αρχή αυτό, ότι στις αρχές ε, Νοεμβρίου θα είναι η ημερομηνία η οποία τελικά θα ισχύσει. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα ισχύει για την Επιτροπή. Ναι, αλλά ελπίζω ότι όλοι μας θα συμπαραταχθούμε και να, θα πρέπει να ζητήσουμε κάποια ελαστικότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να είμαστε πολύ στεναροί και να υποστηρίξουμε με πυγμή αυτή τη θέση. Ορισμένοι συνάδελφοι τάχθηκαν υπέρ μιας νέας στρατηγικής. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσης θα πρέπει να είναι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Το 2008 και το 2009 εγκρίναμε το νέο ενεργειακό πακέτο για τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Έχουμε τη νέα οδηγία για την ασφάλεια εφοδιασμού για το φυσικό αέριο. Έχουμε το κλιματικό πακέτο, είχαμε την οδηγία για τα κτίρια, για την κτηριακή απόδοση ε, ενέργειας. Και μέχρι το 2020 θέλουμε να μειώσουμε την ενεργειακή ζήτηση και να έχουμε όλο και περισσότερες πηγές. Οπότε η πρόκληση για να επιτύχουμε την ενεργειακή ασφάλεια είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουμε τις υφιστάμενες από νομοθετικές διατάξεις και τις ηλυμένες αποφάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη έχουμε εγκρίνει. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα, απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε για να υλοποιήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν τη εφαρμογή υπάρχουν και άλλα 4-5 πολύ σημαντικά θέματα. Το θέμα των υποδομών για παράδειγμα. Και αυτό είναι θέμα εσωτερικής αγοράς και βελτίωση της ασφάλειας. Ε, επίσης ε, αέριο από σχιστολιθικά στρώματα. Η οι Υπουργοί θα συνεδριάσουν τον Ιανουάριο για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά δεν υπάρχει κανένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει την ε, επιρροή του shale gas ό,τι αφορά την αγορά υγροποιημένου αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Σε τρεις εβδομάδες το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτς θα υποβάλει μια τέτοια μελέτη για το shale gas στην Ευρώπη. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη για την αντίληψή μας περί ενεργειακής ασφάλειας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο κύριος Βέμπερ πολύ σωστά τόνισε την ανάγκη προστασίας του καταναλωτή. Θα πρέπει αυτό το σημείο να το διατρανώσουμε στο κείμενο. Και σωστά το επισημαίνουν οι σοσιαλιστές. Επίσης, χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική εσωτερική αγορά. Το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας λείπει αυτή τη στιγμή από την εσωτερική αγορά. Βλέπω εδώ την τροπολογία 95, Royal, Lange και Goebbels, που προτείνουν ουσιαστικά αναβολή όλων των νέων πρωτοβουλειών για την πολιτική ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εκτός και αν είναι λάθος αυτή η τροπολογία ή την παρεξήγησα εγώ. Γιατί πριν το 2018 σημαίνει ότι ούτε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, ούτε στην επόμενη θα έχουμε νέες πρωτοβουλίες. Ενώ υπάρχουν ήδη πολλές ατέλειες στην αγορά σας. Ε, θα παρακαλώ λοιπόν να παραμείνουμε στο αρχικό κείμενο που μιλάει για το 2012 και να μην στήσετε παράταση μέχρι το 2018. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι ούτως ή άλλως σκληρές με τα κράτη-μέλη. Θα υπάρξουν κάποια κονδύλια για την έρευνα αν όμως δώσουμε τα χρήματα που ζητάνε τα προγράμματα, ουσιαστικά θα πρέπει να αφιερώσουμε το 90% του ενεργειακού μας προϋπολογισμού στο πρόγραμμα μόνο ΕΤΑ. Ας μην το ξεχνούμε αυτό. Και τέλος, ο αγαπητός Αλέχο αναφέρθηκε σε ορισμένες ουτοπικές τροπολογίες. Δεν ξέρω αν υπενισόταν τις δικές μας. Αλλά υπάρχουν και τροπολογίες για την ενεργειακή κοινότητα. Η IAA που δεν είναι ακόμη ε, πράσινη οργάνωση, σε ένα από τα σενάρια της μιλάει για 75% ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και το παρουσιάζει ως ρεαλιστικό σενάριο, 35% μέχρι το 2020. Οπότε έχουμε τεράστιο δυναμικό και στη Βόρεια Θάλασσα για αιωλική ενέργεια, παράδειγμα. Οπότε μια ενεργειακή κοινότητα έχει νόημα εφόσον στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα, στη μετάβαση, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και για την πυρηνική ενέργεια έχουμε τη συνθήκη Ευρατόμ. Αν θέλουμε λοιπόν σοβαρά μια ενεργειακή κοινότητα, θα πρέπει να πούμε τι ακριβώς θέλουμε, τι περιμένουμε από αυτή την ενεργειακή κοινότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Μπομπίνσκα, για την ε, εξαιρετική δουλειά της. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ σημαντική έκθεση ε, και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι οι θέσεις και ο ρόλος του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής μας στα θέματα που αφορούν στη νέα ενεργειακή ασφάλεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γίνονται αποδεκτά, ακούγονται και συγκρατούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως από το Συμβούλιο. Ε, να σας ευχηθώ και καλή δύναμη για αυτήν την χιονοστιβάδα τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και που υπογραμμίζουν τη σημασία της έκθεσης ε, που έχετε, το σχέδιο της οποίας μας έχετε παρουσιάσει. Συμφωνώ με την ε, παρατήρηση του συναδέλφου, του κυρίου Βίνταλ Κουάντρας, ότι θα πρέπει να αποφύγουμε εθνοκεντρικές λογικές στην προσέγγιση αυτού του ζητήματος, να αποφύγουμε στην πραγματικότητα ένα λάθος που κάνει συχνά το Συμβούλιο ε, και να αποφύγουμε επίσης ουτοπικές προσεγγίσεις. Ε, θα πρέπει όμως ταυτοχρόνως ε, να συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε φιλόδοξες προσεγγίσεις εφόσον μιλάμε για την στρατηγική, την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την, για την επόμενη δεκαετία. Η νέα ενεργειακή στρατηγική, αυτή που κουβεντιάζουμε, έρχεται σε συνέχεια βεβαίως της προηγούμενης και άρα βασικός στόχος είναι να εντοπίσουμε τις αδυναμίες από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, το επισήμαναν αρκετοί συνάδελφοι αυτό, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και τα λάθη του παρελθόντος και να διαμορφώσουμε φιλόδοξες προτάσεις για το μέλλον στη βάση των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, έτσι όπως αποτυπώνονται πια και στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, ε, δηλαδή ε, για την πρόθεση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ε, προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Εφόσον συμφωνούμε ότι αυτή είναι η στρατηγική ε, στόχη της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και είναι οι στόχοι που μας ενώνουν, νομίζω ότι θα πρέπει οι πολιτικές μας προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία να υπηρετούν ακριβώς του στόχους αυτούς, που σημαίνει να συμβάλλουν στην σταδιακή μείωση, στη σταδιακή απεξάρτησή μας από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή ε, των πολιτικών που εμπεριέχονται στο κλιματικό και το ενεργειακό πακέτο που ψηφίσαμε ε, πρόσφατα. Στη μείωση λοιπόν των συμβατικών καυσίμων που θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και τον περιορισμό της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες. Μια δεύτερη βασική προτεραιότητα είναι η βελτίωση και η διεύρυνση των κοινοτικών πόρων που στοχεύουν ακριβώς στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή, να δώσουμε βαρύτητα στην αναζήτηση νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων ε, για τη χρηματοδότηση ενεργειακών σχεδίων που προάγουν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και τέτοια σχέδια είναι υποδομές. Είπε πρόσφατα ε, ο πρόεδρος Μπαρόζο μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη έκδοση ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών σχεδίων. Τα ενεργειακά ε, σχέδια θα μπορούσαν ασφαλώς να εμπίπτουν στην κατηγορία ε, αυτή. Γενικότερα, εν και της παρουσίασης της ανακοίνωσης της Επιτροπής, για τα ε, δίκτυα ενέργειας. Ε, η τρίτη προτεραιότητά μας σε σχέση με την ε, νέα ενεργειακή στρατηγική πρέπει ασφαλώς να είναι ο εξυγχρονισμός και η αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας και κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστική σημασίας για την προώθηση και για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η προώθηση Τη χρήση ευφυών δικτύων και έξυπνων μετρητών είναι στοιχεία που τα αναφέρει στην έκθεσή της ε, η κυρία Μπομπίνσκα, που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ε, προώθηση ε, του στόχου της ενίσχυσης της, της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τέλος, θέλω να πω σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση της ενέργειας, ότι είναι πολύ βασικό και είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει το Κοινοβούλιο να επιμείνει πολύ, ε, και που ε, το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να επιμείνει πολύ περισσότερο από το Συμβούλιο σε αυτό το σημείο για ευνόητους λόγους, ότι η Ένωση θα πρέπει να αρχίσει να μιλάει με μία φωνή στα ζητήματα της ενέργειας, κυρίως ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση της ενέργειας, τις σχέσεις με τρίτες χώρες ε, και να προωθήσουμε ασφαλώς την πολιτική της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και οδών, χωρίς εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Για να αναφέρω ένα, ένα παράδειγμα, συμφωνούμε για την καθοριστική σημασία του νότιου ε, διαδρόμου. Ε, ας προωθήσουμε από κοινού όλα τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο, νότιο διάδρομο και εκείνο που θα οριμάζει ταχύτερα θα προχωράει πρώτο. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, για παράδειγμα, ναι στο Ναμπούκο, όχι στον ITGI, ε, δεν έχουμε νομίζω την πολυτέλεια αυτή. Όχι λοιπόν στους εσωτερικούς ανταγωνισμούς και όχι στους εξωτερικούς ανταγωνισμούς, στις εξωτερικές αντιπαραθέσεις, για παράδειγμα απέναντι στη Ρωσία. Το δικό μας κίνητρο είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού για την Ένωση. Δεν είναι η αντιπαράθεση με καμία ε, χώρα εφοδιασμού, ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, πολύ περισσότερο ε, με τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Äh, Frau Kollegin Ulskog. It's your turn. Tack så mycket. Eh, jag ber också... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα λίγο καθυστερημένα θα ήθελα να συγχαρώ πάντω θερμά την κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε και έγραψε μια πολύ αξιόλογη έκθεση. Νομίζω ότι έχουμε πια καλές προϋποθέσεις και πρόσφορα έδαφος για να καταλήξουμε σε αρκετές συμβαστικές λύσεις. Κάτι που είναι απαραίτητο αν θέλουμε αποτελέσματα κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα που μας αναπτύσσει πολύ ωραία η κυρία και στην έκθεσή της είναι η ιδέα της ενεργειακής απόδοσης το θέμα της βιωσιμότητας, της ε, προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών, αλλά έχουμε και την ε, κοινωνική διάσταση. Η ενεργειακή απόδοση είναι κάτι συναρπαστικό και νομίζω ότι υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση ως προς την ανάγκη επικέντρωσής μας στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη. Αυτό που μας μένει είναι να πιέσουμε τις ε, χώρες που δεν έχουν ε, λάβει ακόμα σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα να κινητοποιηθούν. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη ενεργειακής απόδοσης παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά να προσελκύσουμε και επενδύσεις στο θέμα αυτό. Ο ρεαλισμός επίσης είναι κάτι απαραίτητο, αλλά πιστεύω ότι η ενεργειακή απόδοση είναι πολύ ρεαλιστικός στόχος. Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση και το θέμα της ε, βιωσιμότητας και της ευφορίας φυσικά θα πρέπει να αποφύγουμε υπερβολικά ουτοπικές ε, απαιτήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι παραδοσιακές συμβατικές πηγές ενέργειας είναι ρεαλιστικές και όλες οι καινούριε είναι εφάνταστες ή ουτοπικές. Θα πρέπει να έχουμε μια μακρόπνοη προοπτική και να υιοθετήσουμε και ένα στρατηγικό σχέδιο, γιατί αυτό το νόημα έχει ε, το στρατηγικό σχέδιο. Δίνει μια μακρόπνοη, μακροπρόθεσμη στρατηγική και προοπτική. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας και να ε, εντατικοποιήσουμε τη χρήση τους. Κάτι που ήταν οτοπικό πριν από 20 χρόνια, όπως ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σήμερα είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Εγώ δεν φοβάμαι τις ουτοπικές προτάσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και να μην εγκλωβιστούμε στη σημερινή πραγματικότητα, να υιοθετήσουμε και μια μελλοντική προσέγγιση, μια, να είμαστε διορατικοί. Ως, προ προς την διαφοροποίηση, φυσικά και θα πρέπει να δοκιμάσουμε και νέες ιδέες, να επενδύσουμε σε νέες μορφές ενέργειες. Το θέμα της ε, προστασίας του καταναλωτή ή η προοπτική του καταναλωτή επίσης είναι σημαντικό για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και το θέμα του ανταγωνισμού είναι πολύ σημαντικό, γιατί ελάχιστη διαφάνεια υπάρχει, ενώ τεράστια κονδύλια διακινούνται στον τομέα αυτό. Και πολύ συχνά τα κράτη-μέλη γίνονται έρμεα ή εχμάλωτοι των πολυεθνικών, γιατί δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτούν καλά τα συμφέροντά τους και να λάβουν καλά αποτελέσματα και συμφέρουσες συμβάσεις με τις ε, μεγάλες εταιρείες. Είναι πολύ σημαντικό να αποκαταστήσουμε μια διαφάνεια στην αγορά της ενέργειας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δημοσιονομικά μέσα με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να υποφεληθεί ο καταναλωτής. Ορισμένοι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμένουν σε περιοχές ή ανήκουν σε στρώματα που χαρακτηρίζονται από ενεργειακή ένδυα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη και πιο δίκαιη κατανομή των ενεργειακών πόρων για να αποφύγουμε αυτή την ανισότητα και να δείξουμε μεγαλύτερη ελληνική και στο θέμα της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα, Δεν είμαι υπέρ της ε, θέσπισης υποχρεωτικών οδηγιών προς τα κράτη-μέλη για το πώς θα πρέπει να διαμορφώνουν το ενεργειακό τους μείγμα. Γιατί με μια τέτοια παρεμβατικότητα ουσιαστικά θα εξωθήσουμε τα κράτη-μέλη σε διαμαρτυρίες. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, πολλές χώρες ε, τη θεωρούν προτεραιότητά τους. Στην πατρίδα μου υπάρχει διαφωνία ακόμη και εντός της Βουλής και είναι πολύ σφοδρή η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Πάντως κρίμα θα ήταν αυτό το, αυτή η πρόταση για δεσμευτικούς στόχους ό,τι αφορά το ενεργειακό πακέτο. Θα ήταν πολύ ατυχές κάτι τέτοιο. Έχουμε και την πυρηνική ενέργεια, έχουμε και άλλες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην διαφοροποίηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ε, πώς θα δημιουργήσουν το ενεργειακό τους μείγμα. Ο κύριος Χένεν. Ε Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, θα ήταν βαρετή συζήτηση αν δεν υπήρχαν διαφωνίε. Όμω συμφωνούμε σε δύο πράγματα. Καταρχά, τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή κοινότητα ε, ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στην αναγκαιότητα ύπαρξη μια νέα στρατηγική. Όμως θα σταματήσουμε στον τίτλο απλώς, ε, γιατί μπορεί να μην συμφωνούμε σε αυτό που θα πρέπει να συμπεριλάβει η νέα αυτή στρατηγική. Οι ενεργειακέ προκλήσει που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά, τις επόμενες, κατά τα επόμενα δέκα ε, χρόνια είναι τεράστιες. Ε, ενεργειακή παροχή ενέργειας ε, σε αξιόπιστου καταναλωτές, χαμηλότερε τιμές, κάτι το οποίο περνάει μέσα από την θέρμανση του πλανήτη, τις τιμές του πετρελαίου κλπ. Όλες αυτές οι προκλήσεις ε, έχουν να κάνουν με την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το θέμα, τα θέματα της ενέργειας. Γιατί ο ανταγωνισμός, η αποδυνάμωση των ολοκληρωμένων ε, ε, στρατηγικών έχουν ως αποτέλεσμα μια κατάσταση που δεν ε, είναι αυτή που θα θέλαμε, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ελεηλασία ορισμένων πόρων χωρίς καμία απολύτως, ε, κανένα απολύτως ε, αποτέλεσμα για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικότερα για ε, την πυρηνική ενέργεια, γιατί δημιουργεί συμπεριφορές απαράδεκτες, οι οποίες ε, μειώνουν την προσφορά για την αύξηση ακριβώς των τιμών και είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να ε, διαιωνίζουμε το, το πρόβλημα. Η έκθεση που συζητούμε σήμερα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε λοιπόν σήμερα ε, αν δεν θέλουμε να καταργήσουμε όλα τα δίκτυα ενέργειας, αν δεν θέλουμε να ανοικοδομήσουμε από την αρχή τον, ε, τον τομέα της ενέργειας ε, και αν δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προκειμένου να μην παραμένουμε μόνο στο lobbying ορισμένων μεγάλων εταιριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, αμοιβαιότητα ε, και συνεργασία ε, μεταξύ των ε, μεγάλων ενεργειακών μονάδων με σκοπό τελικό την ανταπόκριση στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Κύριε Κρούτς, που δεν μπορώ να προφέρω το όνομά σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα, πολύ ωφέλιμα σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση είναι όντω δύσκολη. Ξεκινάει μια συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική μέχρι το έτος 2020 και είναι πραγματικά δύσκολο εγχείρημα το οποίο ανέλαβε η καθηγητρία Κολάσκα Κολάσκα-Πομπίνσκα Και θεωρώ ότι είναι επιτυχές το αποτέλεσμα. Τη συγχαίρω. Καταρχάς να σας πω ότι η βάση για τις σκέψεις αυτές είναι οι διατάξεις περί σε ό,τι αφορά την ανεργία στη συνθήκη της Λισαβόνα. Και επίσης τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πολιτική ενεργειακή θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα βασικό στόχο, τον καταναλωτή, τον χρήστη, τον πολίτη και όταν μιλάμε για τον ενεργειακό τομέα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά ιδιαίτερα τον πολίτη το θέμα αυτό, οι οποίοι φαίνεται ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Γιατί αυτό φυσικά πλήττει ιδιαίτερα για το πρωτοφόλι του πολίτη, αλλά και τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες. Πρόκειται για μένα στενή σύνδεση. Και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να επιστήσω την προσοχή σα στο εξή. Αυτή η έμφαση στη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές πηγές, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ε, προμήθειες και την κατεύθυνση από την οποία έρχονται σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον αγωγό Ναμπούκο και εναλλακτικέ πηγέ. Τα θέματα των εναλλακτικών πηγών είναι ιδιαίτερα σημαντικά και αυτά. Και θα καθορίσουν και τη μελλοντική συζήτηση, καθώς θα θέσουν πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που σημειώνετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων κρατών μελών. Κάποια εξ αυτών βασίζονται στον άνθρακα, κάποια άλλα στην πρινική ενέργεια. Δεν δείχνουμε κάποια προτίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάποια πηγή ενέργειας και είναι σαφές ότι υπάρχουν ε, επικριτές και για όλα, για όλες τις πηγές ενέργειας. Η διαδικασία αναδιαμόρφωση σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ε, πηγές, σε ό,τι αφορά και την υδροελεκτρική ενέργεια, ασφαλώς και θα πάρει κάποιο χρόνο. Αυτό φυσικά πρέπει να τύχει και της κοινωνικής ε, αποδοχής. Χαίρομαι και συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Βιδάλ Αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και στην έκθεση αυτή. Μήπως θα πρέπει να αποφύγουμε τροπολογίες οι οποίες είναι υπερβολικά αισιόδοξε. Ε, να μην τις πω ουτοπικές, αλλά υπερβολικά αισιόδοξε. Να τις αποφύγουμε τις τροπολογίες αυτές, να ε, εστιαστούμε κυρίως σε συγκεκριμένες τροπολογίες και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει το έργο και της κυρίας ε, Μπομπίνσκα. Και φυσικά ο απότερος στόχος θα πρέπει να είναι η κοινή ενεργειακή πολιτική. θα πρέπει να τονίσω ότι είναι πολύ κατάλληλη η χρονική συγκυρία και θα πρέπει να τονίσουμε ότι θέλουμε να συμπεριληφθούν τα συμπεράσματά μας. Σα συγχαίρω κυρία Ποβίνσκα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Να δώσω το λόγο λοιπόν πάλι στην συνάδελφο Κολάσκα Ποβίνσκα για λίγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για τους ενεργειακούς στόχους και το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον μας, η οποία είναι πολύ καλή έκθεση, στην οποία αναφέρονται τέσσερις, πέντε βασικοί στόχοι. Και μπορούμε λοιπόν να δούμε τις συζητήσεις και να τις εστιάσουμε τις συζητήσεις μας στα τα σημεία Διαφωνώ με τον συνάδελφο που είπε ότι μερικές φορές η συμφωνία είναι ανιαρή. Λάθος. Απλώς θα πρέπει να κάνουμε μερικές φορές υποχωρήσεις για να καταλήξουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι έχουμε το πλαίσιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και η σημερινή μας συζήτηση δείχνει ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, άσχετα με την ομάδα από την οποία ε, προερχόμαστε, να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία κοινών στόχων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινή ενεργειακή πολιτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα και αυτό το μήνυμα θα στείλουμε με αυτή τη συζήτηση και με, την, με τις τροπολογίες μας και τις συμβαστικές μας προτάσεις. Γιατί όπως σας είπα είναι τόσες πολλές τροπολογίες που κάθε ουσιαστικά παράγραφος θα είναι καρπός συμβιβαστικών ε, προτάσεων και λύσεων. δεν μιλάμε μόνο για ενεργειακή αλληλεγγύη στην έκθεση. Μας ενδιαφέρουν και τα συμφέροντα του καταναλωτή και η προστασία του καταναλωτή. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα οδεύσουμε στις διάφορες τροπολογίες και συμβαστικές τροπολογίες. Είναι αναφίβολα πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα για μας. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ε, είναι θέμα ενεργειακού μείγματος. Ελπίζω να καταλήξουμε και εδώ σε μια συμβαστική τροπολογία. Παρά τη διαφοροποίηση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς όμως επειδή υπάρχει διαφοροποίηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διστάμενες απόψεις για ορισμένες χώρες που με πολλή δυσκολία και αργό ρυθμό θα προσπαθήσουν να απεξαρτηθοποιηθούν από, τον άνθρακα, θα, πρέπει απέναντί να δείξουμε κάποια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ενεργειακού του σμίγματος. Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση και στην εξωτερική πτυχή της ενεργειακής μας πολιτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπογραμμίζεται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και στη δική μου έκθεση έδωσε έμφαση στο θέμα αυτό, γιατί θέλουμε να υλοποιήσουμε κάποιους στόχους που μέχρι στιγμής δεν τους καταφέραμε. Ένα είδος συνέργειας μεταξύ της εξωτερικής ε, ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και της ε, εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν θέλουμε κοινά δίκτυα και κοινή αγορά ενέργειας, θα πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση και να λάβουμε περισσότερο υπόψη τις εξωτερικές πτυχές μιας τέτοιας ενεργειακής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε και τις συζητήσεις ε, και τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα. Σα ευχαριστούμε και εμείς. Να ήθελα να, να σημειώσω το εξής. Επειδή καθυστερήσαμε, θα πρέπει να βιαστούμε λίγο στη συνέχεια. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ δύο-τρεις ε, παρατηρήσεις, γιατί ο συνάδελφος ε, Τούρμε ανέφερε δικές μου παρατηρήσεις. Αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα, αν και έφυγε τώρα. Η τροπολογία που υπέβαλα δεν μιλάει για την περαιτέρω για την περαιτέρω καθυστέρηση τη εξέλιξη τη έννοια του ανταγωνισμού. Όχι, είναι παρεξήγηση αυτό το θέμα. Είναι πότε θα είναι η σωστή χρονική στιγμή για να ελέγξουμε πώ έχει τροποποιηθεί η κατάσταση, πώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και βλέπω ότι και κάποιοι συνάδελφοι στο τελευταίο πακέτο για τις ενιαίε αγορά είχαμε μια βάση εξέταση, η οποία δεν είχε λάβει υπόψη τη σύγχρονη κατάσταση. Καταρχά, λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν τα όσα έχουν αποφασιστεί, μετά να γίνει ένας έλεγχος της ε, κατάστασης και μετά να γίνει προσαρμογή. Αν ε, αυτά γίνουν το 2011, πώς θα μπορούμε το 2012 να εξετάσουμε το αποτέλεσμα της πολιτικής. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα-δύο χρόνια για να εξαγάγουμε συμπεράσματα και συμπεράσματα. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Την τελευταία φορά ήταν μεγάλη η διαφωνία για το κατά πόσον είχαμε τα πλέον σωστά στοιχεία ως βάση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μια δεύτερη παρατηρήση διευκρινιστική. Θεωρώ ότι όλοι όσοι πήραν το λόγο για την πυρηνική ενέργεια δεν θέλουν να πούν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πυρηνική ενέργεια από όλα τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να προδιαγράψουμε κάτι τέτοιο ούτε μπορούμε να προδιαγράψουμε την ε, χρήση άνθρακα ή ανανεώσιμων ε, ενεργειών. Δεν πρόκειται για θέμα προδιαγραφής. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά για την πυρηνική ενέργεια θεωρώ ότι, τουλάχιστον το είπε και ο συνάδελφος Σιμπόποντα, το θέμα είναι το εξή. Θα πρέπει να επιτρέπεται τα κρατημέλη να τη χρησιμοποιήσουν. Πρόκειται για μία μόνο εναλλακτική λύση. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για προδιαγραφή. Δεν εννοούσε αυτός, ο κύριος Σβόμποντα. Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στο 5, αφού εγκρίναμε και τα πρακτικά. Στο 5 μιλάμε για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την υποπτία της αγοράς. Η συνάδελφος Λάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία ε, τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά ε, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, οπότε θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πλαίσιο του ε, συγκεκριμένου ζητήματος. Πρόκειται για την Οδηγία 95-2001, η οποία θα έπρεπε να αρχίσει να ισχύει από τις αρχές του 2004. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε όμως για αναθεώρηση της οδηγίας και παρουσίασε μία εικόνα της κατάστασης, αναλύοντας μεταξύ άλλων τις βασικές δυσκολίες ε, που διαπιστώθηκαν. Ουσιαστικά η μεταγραφή της οδηγίας 95-2001 από πλευράς κρατών μελών επειδή δίνει τη δυνατότητα ευχέρεια στα κράτη-μέλη ε, δεν έγινε ομοιογενός παντού και επομένως ε, σκοπό, ε, ο σκοπός της αναθεώρησης είναι ένας καλύτερος συντονισμός. Παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα σε σχέση με τους τομείς εφαρμογής της οδηγίας και ειδικότερα σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα επικύρωσης καταρχάς και έχουμε και ένα πρόβλημα εφαρμογής των προδιαγραφών. Έχει πολύ εξελιχθεί η αγορά τα τελευταία χρόνια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη διαβούλευση για να διαπιστώσει κατά πόσο πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Το άρθρο 40 του κανονισμού 765-2001 προβλέπει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία μέχρι το 2000, πρέπει να αρχίσει να ισχύει μέχρι το 2013 η οδηγία περί εποπτείας της αγοράς. Υπάρχει το κριτήριο βάσει του οποίου θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι ασφαλές ή όχι ένα προϊόν, πρόκειται για το άρθρο 3 της οδηγίας, εξηγείται στο άρθρο αυτό πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα ασφαλές προϊόν. Από την άλλη υπάρχει και το θέμα της ε, ε στο άρθρο 5 υπάρχει υποχρέωση από τους παραγωγούς να δίνουν πληροφορίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή να μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την προέλευση του προϊόντος, να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον ίδιο τον παραγωγό, όπως επίσης και τα στοιχεία, ε, τις λεπτομέρειες της ε, παραγωγικής μεθόδου. Υπάρχει επίσης και το άρθρο 11 της οδηγίας που αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που σκοπό έχουν να περιορίσουν την ε, τοποθέτηση του προϊόντος, στην, ε, του, του προϊόντος που κρίνεται μη ασφαλές στην αγορά. Κάτι ακόμη που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα της διαδικασίας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση παρουσίας στην αγορά επικίνδυνων προϊόντων ή λιγότερο ασφαλών. Πρόκειται για το άρθρο 13 της οδηγίας ε, η κατάσταση είναι διαφορετική από το ένα κράτος μέλος στο άλλο επί του θέματος ε, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας είναι απαραίτητη. Πρέπει ε, επίσης ε, να βρούμε λύσεις που να είναι κοινέ, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μπορούν να εργαστούν επί μίας βάσεως. Υπάρχουν βέβαια και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και έχω σκοπό προς αυτή την κατεύθυνση, με αυτό το γνώμο να συντάξω την γνωμοδότησή μου. Η εφαρμογή της εποπτείας ε, της αγοράς ε, είναι ένα... Ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές, μπορούν να έχουν μπορούν να προσφύγουν στο συγκεκριμένο σύστημα για να μπορούν να γνωρίζουν ε, ποια ε, προϊόντα είναι ασφαλή και ποια είναι λιγότερο ασφαλή. Υπάρχει επίσης και το ζήτημα της ε, τυποποίησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει κάποια κριτήρια. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την οποία ήμουν σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚΑ βασίστηκα σε μελέτες ε, στην ανάπτυξη της τυποποίησης ε, και την ε, βελτίωση των διαδικασιών για τις οποίες θεωρεί ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την γενική ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και για την εποπτεία της αγοράς. Θα ήθελα επίσης να σας εκφράσω και κάποιες σκέψεις μου. Ελπίζω να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη, να μην κάνουμε διπλή δουλειά με οδηγίες που δεν είναι ενδεχομένως ίδιες, αλλά πολλές φορές καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Για παράδειγμα, η οδηγία για τα παιχνίδια. Έχει ένα συγκεκριμένο στόχο η συγκεκριμένη οδηγία, αλλά κατά κάποιο τρόπο ε, περιλαμβάνει κάποια στοιχεία της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Οπότε καλό θα ήταν να αποφύγουμε τη δημιουργία σύγχυσης ε, με κείμενα που ασχολούνται με το ίδιο πράγμα και πρέπει παράλληλα να στοχεύουμε και σε, μια, σε, σε απλοποίηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ε, παράγουν προϊόντα που είναι ασφαλή, χωρίς να πρέπει να ε, χωρίς να επιβαρύνουμε περισσότερο οικονομικώς ε, για επιπλέον δοκιμές ε, ασφάλειας των προϊόντων. Κάτι ακόμη που αναφέρθηκε είναι η ανάγκη ύπαρξης πιο ενιαίας νομοθεσίας. Αυτά ήθελα να σας πω στο πλαίσιο της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Ούτω ή άλλω ε, χάσαμε και πολύ χρόνο συζητώντα το πρώτο θέμα τη ημερήσια διάταξη, οπότε καλύτερα να σταματήσω εδώ. Εγώ θα, συζητήσω με, θα συζητήσω με τους κοιόδης εισηγητές και βέβαια ε, θα ε, δούμε πώ θα δω πώ μπορούμε καλύτερα να βελτιώσουμε το κείμενό μα. Σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ που καταβάλλετε και προσπάθεια να είστε πιο σύντομοι. Ο συνάδελφο Μπουτικόφερ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ω κοιόδη εισηγητής εξ ονόματο τη ομάδα μου, θα ήθελα να τονίσω λίγα στοιχεία θεωρούμε ότι βασικά είναι πέντε στοιχεία. Καταρχάς, θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί η εποπτεία της αγοράς επί της ουσίας δεν λειτουργήσε. Σε τι οφείλεται, ποια είναι η αιτία και τι θα πρέπει να κάνουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κατά δεύτερον, μιλήσαμε για ανεξάρτητη αδειοδότηση από τρίτο μέρος. Κατά τρίτον, για την καλύτερη ανιχνευσιμότητα των προϊόντων και των ε, διαδικασιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά επικίνδυνα προϊόντα. Κατά τέταρτον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε την κοινή δήλωση της ΑΝΕΚ και της BUEC σε ό,τι αφορά το θέμα του πώς μπορούμε να δράσουμε πιο γρήγορα όταν υπάρχει κίνδυνος υγείας και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών τυποποίησης και κατά πέμπτον, σε ό,τι αφορά τα θέματα τυποποίησης τα οποία συζητήσαμε, εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μια διαδικασία fast track γρήγορης διεκπαιρέωσης προκειμένου να περιοριστούν χρονικά τέτοιες παραμονές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Εντάξει, ωραία. Έχουμε και άλλες ε, ευκαιρίες να συζητήσουμε. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη λοιπόν για την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συνάδελφο Μαρινέσκου είναι αρμόδιο και του δίνω πάρα αυτό το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τρεις τομείς για τους οποίους θα χρειαστεί να βρούμε καινοτόμο χρηματοδότηση. Οι τομείς είναι οι κλιματικές αλλαγές, η ανάπτυξη και θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα της χρηματοδότησης ε, δίνοντας έμφαση στην οικονομική μεγέθυνση. Γιατί μερικές φορές ε, τα μέσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Η καινοτόμως χρηματοδότηση για το περιβάλλον και την καταπολέμηση των κοινωνικών αλλαγών θα πρέπει να υλοποιούν δύο στόχους. Μέσο και μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονη αύξηση των ε, δημοσίων εσόδων. Θα πρέπει να θεσπίσουμε φορολογικά κίνητρα προκειμένου να, να ενθαρρύνουμε τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει η τρέχουσα ενεργειακή κρίση να μας εξωθήσει στο να σπεύσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις στα προβλήματά μας. Η καινοτόμο χρηματοδότηση για την ενέργεια είναι πολύ σημαντική για να ξεφύγουμε από την σοβούσα ενεργειακή κρίση. Ο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη φορολογία, γιατί η ύπαρξη διαφορετική φορολογία στα κράτη-μέλη ίσω δημιουργήσει στρέβλωση ανταγωνισμού και διατάραξη τη ενιαία αγορά θα πρέπει να βρεθούν κάποια μέσα και για την φορολογία του άνθρακα, αλλά και για συστήματα που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ένα τμήμα των εσόδων που προέρχεται από αυτή την φιλοπεριβαλλοντική φορολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τα μέτρα που στόχο τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και βελτίωση της ενεργειακής υποδομής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και την αναχρησιμοποίηση των αναξιοποίητων κονδυλίων. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν κονδύλια που μένουν ανεκμετάλλευτα. Επίσης, ε, ο φόρος για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα πρέπει να ε, περικόψει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να πλήξει τις επιχειρήσεις. θα πρέπει επίσης να ξεχνούμε τα, αποτελέσ... τα συμφέροντα του καταναλωτή. Προτείνουμε και τη δημιουργία ευρωομολόγων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρόλε. Ευχαριστώ. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ με το σχέδιο γνωμοδότηση του κ. Μαρινέσκου, γιατί είναι εξισορροπημένη και παρουσιάζει τι βασικέ αρχέ τη φορολογία ε, ε, για τον άνθρακα. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με ολόκληρη την ιδέα του φορολογικού συστήματος για τα ορυκτά καύσιμα. Όμως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα ανταγωνισμού που αφορούν ειδικότερα στο θέμα της ε, φορολογίας τέτοιου είδους και πρέπει επίσης να, να, να δούμε πραγματικά το γεγονός ότι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τη φορολογία δεν είναι μόνο κάτι που θέτει νέες αρχές, αλλά είναι και κάτι το ε, ιδιαίτερα προβληματικό. Οι αρχές αυτές δηλαδή είναι προβληματικές και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε κάτι τέτοιο στο Συμβούλιο, το να... Ε, να προβλέψουμε τη διάθεση των, των εσόδων αυτών. Και θα ήθελα επίσης να σχολιάσω το θέμα της ε, οικονομικής σταθερότητας, ε, ε, την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους. Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Έχουμε από τη μία την οικονομική σταθερότητα και από την άλλη τον τρόπο ε, εξέβρεσης ε, ορισμένων επιπλέον ε, πόρων, επιπλέον χρηματοδότησης. Και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε αυτά τα δύο να αναφέρονται στο ίδιο κείμενο. Ευχαριστώ. Miss Ford, excuse me. Thank you very much and thank you. Κυρία Φόρντε, ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και ελπίζω να μπορώ να βοηθήσω την Επιτροπή σας ενημερώνοντας για τις τελευταίες εξελίξεις ε, ε, στην ΕΚΟΝ σε ό,τι αφορά την καινοτόμο χρηματοδότηση. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότηση των υποδομών για τη στρατηγική της για το 2020, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Και επειδή είχα σχετική πείρα και επαγγελματική, είμαι υπέρ της ε, ε, αποτελεσματικής και καινοτόμου χρήσης ε, και των κρατικών κονδυλίων αλλά και των ιδιωτικών κονδυλίων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν υποδομές και να γίνουν επενδύσεις. Χθες στην Επιτροπή Εκών είχαμε δημόσια ακρόαση με την ΕΤΕ και αναλύσαμε και το θέμα των ευρωομολόγων, που ήταν μια πρόταση Μπαρόζο. Πάντω η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε αντί να χρησιμοποιείται λιγότερο από 1% του κοινοτικού προπολογισμού ε, για τα χρηματοοικονομικά μέσα, να χρησιμοποιείται έω και 20%. Και θεωρούν ότι η χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων και σχεδίων υποδομή ε, είναι πολύ σημαντική και μάλιστα η ΕΤΕ θα χρησιμοποιήσει και δημόσια κονδύλια, κρατικά κονδύλια, ίσως και κρατικά ομόλογα, για να ενθαρρύνει ιδιωτικούς επενδυτές να συμμετέχουν στην ε, χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών. Υπάρχουν διάφορα μέσα για να προσελκυθούν αυτοί οι ιδιώτες, όπως εγγυήσει, για παράδειγμα, αλλά δυστυχώ η κατάχρηση τέτοιων εγγυήσεων και τέτοιων ειδικών ε, χρηματοοικονομικών μηχανισμών είναι που μας οδήγησε στην παρούσα οικονομική κρίση. Θα πρέπει φυσικά να θαρρύνουμε τη χρήση και κρατική, αλλά και ιδιωτική ε, επένδυσης σε καινοτόμου ε, τρόπους χρηματοδότηση, αλλά να μην ξεχνούμε και τον έλεγχο που είναι απαραίτητος. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην διαφάνεια, στις σωστές επενδυτικές οδηγίες, στην αποφυγή της κακοδιαχείρισης, ε, σημαντικό έλεγχο και επίσης ε, λογοδοσία. Γιατί δεν είναι λογικό να μην ε, γίνεται εμβριθής διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για παράδειγμα. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να ακούγεται τη φωνή του. Φυσικά θα πρέπει να ακούμε και το, τη γνώμη των ενδιαφερομένων για θέματα επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τα μόρια για τα, τον άνθρακα, εμείς δεν είμαστε υπέρ ενός ε, πανευρωπαϊκού φόρου άνθρακα. Προτιμούμε τους εθνικούς ε, φόρους, γιατί το θέμα αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Τούν άλλοι τέσσερις συνάδελφοι του λόγου. Θα μπορούσατε παρακαλώ όλοι να είστε λίγο πιο σύντομοι, γιατί θέλουμε να κοιτάξουμε για τα άλλα θέματα. Κύριε Σουζαντό. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στο συνάδελφο Μαρινέσκο για το σχέδιο γνωμοδότησης. Μερικά σχόλια. Εμείς ε, συμφωνούμε με τον εισηγητή όταν λέει ότι πρέπει να επεκτείνουμε τη φορολογία για τον άνθρακα, ε, ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να βρούμε όμως τη σωστή ισορροπία, η εναρμόνιση για το θέμα αυτό είναι ώστό. Πρέπει να, να παρεμποδίζει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν ε, αν θέλουν να πρωτοσταθήσουν επί του θέματος αυτού. Αν υπάρχει, αν υπάρχει εναρμόνιση, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις, ε, να υποβάλουμε κάποιε τροπολογίες για την αναθεώρηση τη οδηγία ε, για τη φορολόγηση της ενέργειας, ε, αλλάζοντα λιγάκι το περιεχόμενο, θέτοντα μία πτυχή για τον άνθρακα, να μπορούμε να αναφερθούμε στο θέμα της επιπλέον χρηματοδότησης όσον αφορά την εμπορία εκπομπών αερίων. Θα ήθελα να, να το επενθυμίσω, αλλά ούτως ή άλλως αναφέρεται στο έγγραφο. Όταν μιλάμε για τη δημοπρασία των ποσοστώσεων υπάρχει το ζήτημα των δωρεάν των δωρεάν κατανομών ποσοστώσεων. Να υπάρξει δηλαδή ένας μηχανισμός, ε, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, που από τη μία θα επιτρέπει τη διαχείριση των πόρων και από την άλλη την προστασία ε, των ευρωπαϊκών εταιριών, ειδικότερα αν κινδυνεύουν λόγω των κλιματικών φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει και το θέμα των μη δαπανών στο ζήτημα αυτών των καινοτόμων, της τόμου χρηματοδότησης, ε, για παράδειγμα ε, ενέργεια από ορυκτά ε, καύσιμα. Δεν είναι κάτι που το ζητά μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το G8 είναι, το, το ζήτησε επίσης. Ε, πολύ καλή ιδέα είναι να ε, συμμετέχουν ε, και οι αεροπορικές εταιρείες στο σύστημα των ποσοστώσεων γιατί θα αυξηθούν έτσι οι δημοπρασίες είτε στο πλαίσιο της εμπορίας εκπομπών αερίων είτε σε επίπεδο διεθνών συμφωνιών. Το να συμπεριλάβουμε επίσης και τις θαλάσσιες μεταφορές είναι κάτι που θα μπορούσε να μας επιφέρει επιπλέον χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα υποβάλουμε και σχετικές τροπολογίες. tänan arvamuse Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συντάκτη γνωμοδότηση για τις πολύ καλέ του προτάσεις. Συμφωνώ με τις περισσότερες, αλλά θα καταθέσω και δικέ μου. Στην πολιτική μου ομάδα εξετάσαμε το θέμα του φόρου άνθρακα και καλό θα είναι να Υποβάλλει πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έκθεση για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου φόρου και μετά να καταθέσει προτάσεις για πανευρωπαϊκή φορολογία άνθρακα. Τα διάφορα φορολογικά συστήματα δεν θα πρέπει να αλληλοαποκλείονται και το κλιματικό πακέτο που ε, υιοθετήσαμε το 2008 προβλέπει ένα καταμερισμό των προσπαθειών και την ανάληψη υποχρεώσεων από όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να υλοποιηθεί ο κοινό στόχος. Ένας πανευρωπαϊκός φόρος άνθρακα ίσως επιτρέψει τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και αν έχουμε μια συντονισμένη κοινοτική προσπάθεια και μια σταδιακή ένταξη της αρχή ορυπαίνων πληρώνει, θα μπορέσουμε και στο μέλλον να περικόψουμε άλλους φόρους, να μειώσουμε το εργασιακό κόστος και άρα να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρινέσκο ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια συντονισμένη προσπάθεια. Αυτή είναι η εποφελέστερη προσπάθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει όμως να τιμωρούμε ουσιαστικά τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη αναλάβει δικές τους πρωτοβουλίες ή να τα φέρουμε σε δυσμένη θέση. Η... Τα περιβαλλοντικά ευρωομόλογα ίσως είναι μια λύση για να καλύψουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε την πρόταση και των Ευρωπαϊκών Πράσινων Τραπεζών. Έχω και άλλες προτάσεις που θα καταθέσω για καινοτόμο χρηματοδότηση. Thank you, Mr. Chair. Firstly, I want to say I'm not a member. Ο συνάδελφος Κέλλη, να πω καταρχάς ότι δεν είμαι μόνιμο μέλος, είμαι αναπληρωτής, αλλά χαίρομαι που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να είμαι μέλος, ωστόσο και θα έπρεπε να είμαι και μέλος. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μαρινέσκου για την έκθεση και για τα σχόλιά του. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ καλή. Και βασικά εδώ πέρα η λέξη κλειδί είναι η καινοτόμος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στα, στον ίδιο δρόμο με του ίδιου τρόπου που είχαμε παλιότερα. Θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση και θα πρέπει πολλά πράγματα να κάνουμε. Καταρχά, θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη και του πολίτε εν γέννη ότι είναι επιθυμητό, θεμητό να υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά μέτρα τα υπάρχουν τα οποία θα πρέπει να τύχουν της ε, υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάπτυξη των δικτύων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όλα αυτά εν ώψη και της ύφεσης και όσο μας δίδαξε η νέα χρηματοδο... η νέα... το νέο τραπεζικό σύστημα και το καθεξής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα καλωσορίσουμε. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές και χειρό το μήνυμα ότι το 0,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάτι να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα όπως είπε ο κ. Μαρινέσκου, με την ιδέα του ευρωομολόγου, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα τύχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν και ελπίζουμε να επιταχυνθεί και η κατάρτιση του σχεδίου, αλλά και η εφαρμογή του σχεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ρουμπίχη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χρηματοδότηση σε εποχές όπως η σημερινή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μαρινέσκου γιατί θεωρώ ότι επί της ουσία ήταν πολύ σωστή η έκθεση του. Ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά τον πληστηριασμό του διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει τα αποτελέσματα, τα έσοδα του πληστηριασμού να διοχετευθούν προς τους σωστούς στόχους και ο πληστηριασμός θα πρέπει να εξυπηρετεί καταρχάς τη βιομηχανία. Είναι σημαντικό λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη σε ό,τι αφορά την φορολογία του τελικού χρήστη, γιατί στην περίπτωση αυτή θα πληρώνουν όλοι και έτσι θα είναι και πάλι ανταγωνιστική η βιομηχανία μας. Άρα, τάσσομαι υπέρ μιας περιορισμένης φορολογίας του τελικού χρήστη. Και αυτό θα συμβάλλει στην αγωνιστικότητα της Ένωσης. Δεύτερο σημείο, φυσικά, υπάρχει και ο φόρος των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούν να καταστούν πιο διαφανή τα παράγωγα και νομίζω ότι θα έπρεπε να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην σταθεροποίηση των αγορών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αύριο θα μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και θα υποχρεωθούμε να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση και για τη χρηματοδότηση της καινοτομία. Είναι και το ζήτημα που συζητούμε αυτή τη στιγμή και είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας προπολογισμό που δεν αυξάνεται ε, ε, αλλά πρέπει γι' αυτό να ορίσουμε προτεραιότητες. Πρέπει να είμαστε δηλαδή καινοτόμοι και στον τομέα της χρηματοδότηση, να είμαστε συνεπεί ε, και αυτό το ή άλλως αναφέρεται και ε, στις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση δεν μπορεί να γίνει διαχείριση σε εθνικό επίπεδο γιατί τότε ε, θα υπησέρχονταν ε, ανισότητες και δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή ε, βιομηχανική πολιτική αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της χρηματοδότησης. Όμως πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα προγράμματα, ο προβληματισμός ε, για τη φορολόγηση του ε, άνθρακα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει να υποχρεώσουμε νομίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει προτάσεις από αυτού. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, χρειαζόμαστε μία πολιτική αμοιβαιότητας γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μείωση, μέτρα μείωσης ε, του άνθρακα. Πρέπει τα μέτρα αυτά να λαμβάνονται σε διεθνέ επίπεδο. Αν μόνο εμείς τα κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε πάντοτε προβλήματα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας οικονομίας μα Γι' αυτό ακριβώς η πολιτική της αμοιβαιότητα, η οποία μπορεί να προβλέψει βέβαια και έναν μηχανισμό ενσωμάτωσης ε, ε, του, του άνθρακα, ε, πρέπει να διερευνηθεί και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ε, ε, δίωδοι, υπάρχουν πολλοί τρόποι, υπάρχει μια πραγματική σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως επίσης και με την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρινέσκο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα σχόλια. Ευχαριστώ καταρχήν τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Ένα σύντομο σχόλιο για το earmarking για την προσημείωση των κονδυλίων. Σίγουρα θα γίνει σφοδρή συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί πολλές χώρες προτιμούν να έχουν τα κονδύλια στον προϋπολογισμό και να τα δια... κατανέμουν κατά βούληση, όχι με προκαθορισμό του προορισμού τους. Θα σας δώσω όμως ένα παράδειγμα. Αν επιβάλλουμε φόρο για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, για τα αεροσκάφη για παράδειγμα, δεν είναι σωστό ένα τμήμα των κονδυλίων αυτών να τα, να τα αφιερώσουμε στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη των νέων κινητήρων που θα ε- εκπέμπουν λιγότερα αέρα θερμοκηπίου. Νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι είναι λογικό κάτι τέτοιο. Ελπίζω να συμφωνείτε και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα τα λάβω υπόψη στην γραμμοδότησή μου. Ευχαριστώ ενημερωτικά να πω το εξή ότι η 12η Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στο 7 της ημερήσιας διάταξης. Μιλάμε για το θέμα το διάσημο πλέμα, πλέον. Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοκρατίας της Κορέας και ο κ. Ντανίλ Κασπάρη είναι ο αρμόδιος για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το έτος 2007 το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συνάψει συμφωνία με την ε, Κορέα. Διήρκεσαν δύο χρόνια οι συναλλαγές, οι διαπραγματεύσεις αυτές και συμφωνία με γραφή στις 15 Οκτωβρίου του 2009. Η συμφωνία θα πρέπει ως πρώτη εμπορική συμφωνία να ε, έχει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω ότι πρόκειται μια τεράστια πηγή ε, ανάπτυξης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλες οι επιχειρήσεις εξαγωγής αποτελούν περίπου το 10% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ορισμένες περιοχές εκπροσωπούν και αν το 50% των εξαγωγών. Θεωρώ ότι θα επωφεληθούν αμοιβαία και οι δύο εταίροι. Θα αυξηθεί η παραγωγή στην Κορέα και θα αυξηθούν κατά 82% οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στην ε, Κορέα. Το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 38% όταν θα καταργηθούν τα δασμολογικά εμπόδια. Οι εξαγωγές μηχανικών και γυρικών προϊόντων προς την Κορέα θα απαλλάσσονται από φόρους έως 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος και σημαντικό νέο εμπόριο θα προκύψει σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους έως 19,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν είναι και γενικά θετική η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζονται θέματα χημικών, ε, φαρμακευτικών προϊόντων και οι αρμόδιες ε, επιτροπές τάχθηκαν υπέρ της ε, συμφωνίας. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα Γι' αυτό προβλέπεται και μερία ρήτρα διασφάλισης για να ανταποκριθούμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες αυτές, για παράδειγμα. σε περίπτωση υπερβολικών εξαγωγών από την Χερσόνησο, την Κορεατική προς την Ευρώπη, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο μηχανισμός ε, ασφάλειας και σύμφωνο και μετά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του αρμοδίου εισηγητή. Θεωρώ ότι έχουμε απευθυνθεί, έχουμε πραγματευτεί τα πιο σημαντικά θέματα τώρα. Πρέπει να επικυρωθεί η συμφωνία και συστήνω να επικυρωθεί. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θα το συζητάμε σήμερα, αλλά θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το θέμα της ρήτρας διασφάλισης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση. Υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου η οποία αποτελεί βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ, Κοινοβουλίου, μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής και ελπίζω να μπορέσουμε να επικυρώσουμε τη, συνθήκη, τη σύμβαση φέτος. Ευχαριστώ, κύριο Σκέλη. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κάσπαρη για την ε, έκθεση του και την γραμματότηση του μάλλον είπε θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και η γεωργία και η βιομηχανία από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ωραία, αλλά ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα για τη γεωργία από το ευρωπαϊκό ε, πρίσμα, γιατί είναι επίμαχο αυτό το θέμα. Μπορείτε να εξασφαλίσετε την ισορροπημένη λήψη υπόψη και της Γεωργίας ό,τι αφορά την απολαβή ε, ωφελών από την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συνεργών με την Κορέα και να μην επικεντρωθούμε μόνο στη βιομηχανία. Ο κύριος Μαρινέσκου. Συμφωνώ με τον κύριο Κάσπαρη και συμφωνώ και με το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή ελεύθερων συναλλαγών πυροδότησε πολλές συζητήσεις, ιδιαίτερα με την αυτοκινητοβιομηχανία. Βέβαια, δεν έχουμε δυνατότητα επιρροής ή τροποποίησης αυτής της συμφωνίας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη δεχτούμε ή να την απορρίψουμε. Πάντως θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπογραμμίσουμε την ανάγκη θέσπισης ενός μηχανισμού που θα εξασφαλίζει προστασία της βιομηχανίας μας σε περίπτωση που οι εισαγωγέ σε ορισμένους κλάδους ε, θα αυξάνονται υπέρμετρα, ιδιαίτερα για τα μικρά οχήματα. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας διαβεβαιώσει ότι ο κανονισμός για το διοξίδι του άνθρακα που ισχύει στην Κορέα δεν θα επιβάλλει ε, μεγάλους περιορισμούς ή επιπλέον υποχρεώσεις στους ε, εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για τα αυτοκίνητα, για να μην δημιουργηθεί έτσι ένας ε, μη εμπορικός φραγμός για το εμπόριο μέσω αυτού του κανονισμού διοξιδίου του άνθρακα της Κορέας. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΗΠΑ και Κορέας. Ας μην ξεχνούμε ότι ό,τι πλεονεκτήματα θα λάβουν οι Ηνωμένες κατόπιν θα μπορούσαν να τα διεκδικήσουν και ε, τα διεκδικήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κορέα. Κυρία Φόρτ, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία μια ολόκληρη σειρά αντίστοιχων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που θα ακολουθήσουν. Και συμφωνώ ότι θα είναι πολλά τα ωφέλη από τη συμφωνία αυτή, αλλά θα πρέπει να είναι όντω συνολική και να μην βρεθούμε σε δυσμενή θέση σε σχέση με τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά να διεκδικήσουμε και εμεί αντίστοιχα ωφέλη. Είναι περίεργο που η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απλώ συμβουλευτική και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε να τροποποιήσουμε τη συμφωνία. Ο κύριος Στάρντι όμως, που είναι ο αρμόδιος για την έκθεση στην ΙΝΤΑ, είπε ότι υπάρχουν πολλά εχέγγυα και ασφαλιστικές δικλείδες για τη βιομηχανία. Και υπάρχει το θέμα του duty drawback, που μπορεί να ωφελήσει οικονομικά που θέλουν να μεταθέσουν την παραγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει τέτοιου είδους περιπτώσεις να λαμβάνουν ωφέλη από δασμούς. Προσοχή όχι μόνο στους ε, δασμολογικούς φραγμούς, αλλά και στους ε, μη δασμολογικούς φραγμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσέξει τις ε, ασφαλιστικές δικλίδες και οτιδήποτε τέτοιο σημείο θα πρέπει να ελέγχεται και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, όχι μόνο τώρα, αλλά και για τις μελλοντικέ συμφωνίες. Ο συνάδελφος Κασπάρη, να απαντήσω στις ερωτήσεις πολύ γρήγορα. Μιλήσατε για τη Γεωργία, για παράδειγμα. Είναι δραματικές, ε, μάλλον τεράστιε οι μειώσει των δασμών στον τομέα αυτό. Σε κάποιους τομείς ε, καταργούνται τελείω. Ένα παράδειγμα, από την ημέρα σε θέση σε ισχύ της ε, Συμφωνία θα μειωθεί σε μηδενικό συντελεστή η δασμή για το αλκοόλ και έχοντα υπόψη μου την Ιρλανδία για παράδειγμα αλλά και άλλου παραγωγού ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα Ίνου κατά δεύτερον ναι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα στη συμφωνία αυτή μπορούμε να συμφωνήσουμε να διαφωνήσουμε αλλά να σα πω το εξή. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει, δεν υπήρχε ακόμα η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν είχαμε συναπόφαση πολιτικά από πολιτικής άποψης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την αρχή των διαπραγματεύσεων είχαμε εγκρίνει μία έκθεση για την ε, Νότιο Κορέα και είχαμε τοποθετηθεί αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις και κοιτώντας σήμερα το κείμενο του συμφωνίας και το ψήφισμα τότε και το κείμενο του ψηφίσματος βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται το, η συμφωνία σε όλα τα σημεία που θύχθησαν τότε ε, στην, ε, στο ψήφισμα. Και κάτι άλλο για τα προστατευτικά μέτρα τώρα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε για τα προστατευτικά μέτρα στην πρώτη ανάγνωση είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό αφορά και την αυτοκίνητο βιομηχανία και τα μικρά οχήματα. Σε περίπτωση που υπάρξει πλημμύρα, όπως είπα, ε, εισαγωγών στον τομέα αυτό, θα υπάρχουν προστατευτικά μέτρα. Και υπάρχουν και άλλες δυνατότητες ε, υποστήριξης σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουν λάβει σχετικές ε, δεσμεύσεις ε, οι Κορεάτες. Δεν πρόκειται να θέσουν ε, νέα δασμολογικά εμπόδια. Αυτά συμφωνήθηκαν και κατά τις διαπραγματεύσεις. Εγώ θεωρώ ως Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι διεξάγονται πολύ έντονες συζητήσεις με την Κορέα γιατί ξέρει και η Κορέα πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και το Συμβούλιο αποφάσισε μετά από τελικές πιέσει, να μην ξεκινήσει η εφαρμογή τη συμφωνία απο από 1η Ιανουαρίου του επομενου ετου έτους, αλλά από 1η Ιουνίου. Αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μισό χρόνο παραπάνω, να εξετάσουμε και την πλευρά τη Κορέα, να δούμε τι γίνεται και με το σχέδιο για τη ρυθμίση του άνθρακα Νομίζω ότι οι Κορεάτες έχουν καταλάβει ότι ασκούμε πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό λοιπόν θα αποτελέσει το βασικό θέμα. Το έχουν καταλάβει οι Κορεάτες αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν συστήνει η Επιτροπή να περάσει αυτή η έκθεση, να εγκριθεί αυτή η συμφωνία και να προσπαθήσουμε να τεθούν σε εφαρμογή παράλληλα με τη συμφωνία και οι μηχανισμοί ε, προστασίας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ζητά κανείς άλλο το λόγο. Εξαιρετικά. Προσώ ολοταχώς. Και περνάμε στο 8. Θέλαμε να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για την ε, αντιπροσωπεία στο 5ο Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου 16 έως 17 Σεπτεμβρίου στο News, Η συνάδελφο Στράουτμαν ήταν ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας και ε, σύντομα θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό, αν παρευρίσκεται κιόλα. Δεν ξέρω μήπως έχει... Έρχεται. Να την περιμένουμε λίγα λεπτά. Ist auch schön. Machen wir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 Bienvenue. Et euh, nous sommes, nous sommes quelque intéressés, nous sommes intéressés, c'est correct, oui, intéressés euh, de savoir que vous avez. Κύριε Τροτμάν, περιμένουμε πώς και πώς την ενημέρωσή σας α, για την αντιπροσωπεία στο Βίλνιος. Θα τα πω στα γερμανικά. Να μας πείτε, κυρία Γκροστέτ, τι έχετε να μας πείτε για την διακυβέρνηση στο Βίλνις. Μα είναι πολύ πιο όμορφα τα πράγματα στα γερμανικά. Ευχαριστώ. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά ήμουν σε συνάντηση με του ε, Ρωμανους συναδέλφου για θέματα και προβλήματα τύπου. Θα σα κάνω μια σύντομη ενημέρωση για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που μετέβει στο Βίλνιους και μάλιστα με πολυμελέστερη αντιπροσωπεία από άλλε χρονιές. Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου είχε ξεκινήσει στην Αθήνα σε μια συμβολική για τη δημοκρατία ευρωπαϊκή πόλη και ολοκληρώθηκε η πενταετία που είχε προβλεφθεί αρχικά για να δοκιμαστεί αυτός ο νέος τρόπος διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν την πρόσβαση, την ασφάλεια, την ανάπτυξη στο διαδίκτυο. Οπότε το πέμπτο φόρουμ στο Βίλνιους είχε και συμβολικό χαρακτήρα αλλά και μεγάλη σημασία. Ε, Δεκαστήγιο, Μαδουρέλ, Φρανσίσκο Βέγνερ, Βανίστα Ρόι, Σαμπίν Βεράιεν, ε, Μπαντία Κουτσέτ, Μπαλτσίτης, Φιν και Μάριαν Σάκερ ήταν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν σε αυτή την ε, αντιπροσωπεία. Είχαμε αρκετές διμερείς συναντήσεις κοινοβουλευτικέ με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα του Διαδικτύου. Συζητήσαμε για το ρόλο αυτού του Ιδρύματος που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τις ε, κοινοβουλευτικές οργανώσεις και τις ομάδες εργασίας που μαζί με εμπειρογνώμονες από επιχειρήσεις και οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών ασχολούνται με το θέμα αυτό. Είχαμε συναντήσεις και με, κοινοβουλε... και με από την Κένια, Τανζανία και Ουγκάντα. Γιατί στην Κένια θα γίνει το επόμενο φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Γι' αυτό και πέρυσι εγκαινιάσαμε συνεργασία με χώρες της Αφρικής, με βουλευτές από τις αφρικανικές χώρες, για την αντιμετώπιση και συζήτηση κοινών θεμάτων. με τους Λιθουανούς ε, συναδέλφους, αλλά και με αίτημα των ε, Ανατολικοαφρικανών συναδέλφων, ασχοληθήκαμε το θέμα της ε, πολυγλωσίας και τα συναφή ζητήματα. Συναντηθήκαμε και με Βρετανούς συναδέλφους, με τον κύριο Βέρβευ, τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον εκπρόσωπο της κυρία Μάρστρομ, τον Πολωνό Υπουργό Επικοινωνίας για να ετοιμαστεί και η Πολωνική Προεδρία του δεύτερου εξάμεινου του 2011 και εκπροσώπους από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις και με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το φόρουμ της, ε, του ΟΗΕ που θα συνεχίσει αυτό το πέμπτο φόρουμ, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, Επιτρόπου Ρέντινγκ αλλά και μέσω του, της έκθεσής μας ε, για το θέμα αυτό αλλά και το, τη συνεργασία του Συμβουλίου σημειώνουμε πρόοδος ότι αφορά τη θεσμοποίηση θεσμοθέτηση αυτού του φόρουμ που θα γίνει ένα είδος ε, δεύτερου φόρουμ ε, των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θέλουμε όμως επικάλυψη, θέλουμε μια ελαστική οργάνωση. Μια τέτοια απόφαση συνέχισης, αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση συνέχισης αυτού του φόρουμ, το επόμενο φόρουμ θα γίνει στο Ναϊρόμπι. Οι συζητήσει που έχουμε στο φόρουμ αυτό είναι παρόμοιες με αυτές του Κοινοβουλίου, δηλαδή προστασία των παιδιών στο ίντερνετ ασφάλεια και καταπολέμηση του εγκλήματος, πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε στο φόρουμ είναι το cloud computing. Επίσης, η ελευθερία έκφρασης, ε, η... το θέμα του αλφαβητισμού σε θέματα πληροφορικής, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Η Μαρία Μπαντία Κουτσέτ έλαβε το λόγο εκπροσωπώντας την αντιπροσωπεία στο δεύτερο τμήμα. Ε, εγώ ήμουν συντονίστρια στο πρώτο τμήμα και στο δεύτερο συντονίστρια ο κύριος Κάρκλινς, ένας από τους ε, βασικούς διευθυντές της UNESCO. Επίσης μιλήσαμε για το ραδιοελεκτρικό φάσμα, την διαλειτουργικότητα, και για όλα αυτά τα θέματα θα είναι ενδιαφέρον στην πορεία των συζητήσεών μας να περιλάβουμε και τις συζητήσεις και ό,τι προσπαθήσαμε να πάρουμε από το φόρουμ. Θα ήθελα να εκφράζω τις ευχαριστίες μου για όλους όσους συμμετείχαν στο φόρουμ αυτό, στον άμεσο συνομιλητή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ενρίκο Φόρτη, αλλά και το επιτελείο του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο την κυρία Κρούς. Στο μέλλον, αν θέλουμε να έχουμε σημαντικότερη επιρροή σε αυτά τα αιτήσια φόρουμ, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας. Ήταν κάπως παράδοξο ότι ενώ η παρουσία των Ευρωπαίων ήταν πολύ σημαντική, οι Αμερικανοί έλαψαν τη της απουσίας τους. Ε, από πλευρά Ευρώπης είχαμε Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Αλλά χρειαζόμαστε και εκπροσώπους από τη βιομηχανία και από το διπλωματικό κόσμο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις μελλοντικέ διοργανώσεις. Και επίσης θα πρέπει να εμπλακούμε στο δίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης που ονομάζεται Eurodic και να δραστηριοποιηθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Είπαμε στην Επίτροπο Κρούς ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμειχθεί ενεργά. Προτείναμε μάλιστα και προφορική ερώτηση με συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν παγκοσμίω και θέματα που είναι ιδιαίτερα προσφυλή στη δική μας Επιτροπή Βιομηχανίας και που, έχουν, που είναι επίκαιρα, όπως είναι η ουδετερότητα στο διαδίκτυο, το cloud computing, το, το φάσμα κτλ. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και για μας αλλά και για τον κλάδο. Σας ευχαριστούμε κυρία Τροτμάν. Υπάρχουν ερωτήσεις. Όχι, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Στην συνεδρία των συντονιστών που θα ακολουθήσει θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αυτά ως προς την τακτική μας συνεδρίαση. Σε δύο λεπτά θα συνεχίσουμε και κλεισμένο το θυρών οι συντονιστές.